Mes chers collègues, nous allons... Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Mes chers collègues, la commission transport τη συνάδελφοι, Επιτροπή Μεταφορών οργανώνει σήμερα δημόσια Κρόαση με θέμα τον αντίκτυπο του Brexit ε, στην αεροπλοεία. Στόχος της ακρόασης αυτής είναι να ακούσουμε τους εκπροσώπους ε, ξέχοντας εκπροσώπους των αερολιμένων, των αερομεταφορέων ε, της Airbus για το Brexit. Έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα πώς εκτιμούν οι θύνοντες ε, της αεροπορίας το Brexit, πώς βλέπουν το μέλλον και τι έχουν ήδη εντοπίσει από βασικές επιπτώσεις μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι στη δική μας Επιτροπή ασχολούμαστε και με την οικονομική ευρωστία των αερομεταφορέων, μας ενδιαφέρει αυτό, η επίπτωση στην απασχόληση και ε, ενδιαφέρουν επίσης οι εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθούν οι ε, συνδέσεις και η ελευθερία των κινήσεων των Ευρωπαίων πολιτών. Για τον λόγο αυτό, θελήσαμε να διοργανώσουμε τον παρόντο διάλογο, επικοδομητικό διάλογο με τους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες. Είμαστε στο ρόλο μας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας αρέσει να κάνουμε συζητήσεις ουσίας με ειλικρίνεια, με διαφάνεια, έτσι ώστε να αρθούν κάποιες ανασφάλειες που συνδέονται με το Brexit. Διότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ένα κράτος μέλος επιλέγει να μας εγκαταλείψει. Για το λόγο αυτό η παρούσα ακρόαση είναι η πρώτη μόνο από μια σειρά τεσσάρων μεγάλων ακροάσεων. Ο νησιωτικός χαρακτήρας του Ηνωμένου Βασιλείου επιτάσσει να ασχοληθούμε και με την ναυτιλία, εκτός από την αεροπλοεία. Το ίδιο ισχύει και με τις χερσαίες μεταφορές, είτε πρόκειται για οδικές είτε για σιδηροδρομικές. Και η τέταρτη ακρόαση θα είναι αφιερωμένη στους προσώπους του προσωπικού και των επιβατών από κάθε ε, μέσο μεταφοράς που καλύπτει η Επιτροπή μας. Αυτό ήταν το γενικό πνεύμα που πριν τα ανέβει στην Επιτροπή μας. Για την παρούσα τώρα ακρόαση έχω να σας πω τα εξής. Έχουμε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα ακούσουμε τους επικεφαλής τριών μεγάλων αερολιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Heathrow του Λονδίνου, Charles de Gaulle στο Παρίσι και το αεροδρόμιο του Δουβλίνου. Έχουν τις ιδιαιτερότητες τους και τα τρία. το δεύτερο μέρος θα αφιερωθεί στη συζήτηση με τους εκπροσώπους φόρων αερομεταφορέων και τουριστικών επιχειρήσεων. IAG, Ryanair, Airlines for America, Όμιλος Lufthansa ή Όμιλος Τούι. Θα ακούσουμε επίση την εκπρόσωπο της Ερμπά. Μετά από κάθε θα έχουμε και συζήτηση με τους ευρωβουλευτέ. Θα ακούσουμε πρώτα φυσικά τους εκπροσώπους των αεροδρομίων και θα ακολουθεί συζήτηση και στη συνέχεια θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της ακρόασής μας με τους αερομεταφορεί θυμίζω ένα βασικό και πρωταρχικό κανόνα για τη συζήτηση. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα πρέπει οπωσδήποτε να είστε σύντομοι και να εστιάσετε ακριβώς στον αντίκτυπο του Brexit. Σας γνωρίζουμε, γνωρίζουμε το τομέα δραστηριοτήτων σας. Αυτό που σας ζητούμε είναι να αφιερωθείτε σήμερα σε θέματα αντικτύπου του Brexit. Τούτων όλων λεχθέντων σας καλωσορίζω θερμά στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να ανταλλάξουμε απόψεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Επειδή είστε και πολλοί, <laughs> ήθελα να σας πω ότι καλό θα ήταν να περιοριστείτε στα 5 με 7 λεπτά στις ε, παρεμβάσεις σας. Και για όσοι με γνωρίζουν ε, στην Επιτροπή μας, εγώ ορίζω το χρόνο. Θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο ε, στον κύριο Τζον Χόλαντ Κέι. Δεν σας βλέπω. Α, να σας παρουσιάσω. Είστε επικεφαλής του αεροδρομίου του Χήθρο. Ευχαριστώ και καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας. Λέγομαι John Holland K CEO του Heathrow και είμαι και μέλος της ACI Europe, 500 αερολιμένες. Ε, θα σας παρουσιάσω μια κοινή θέση. Είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο Καταρχάς πιστεύω ότι η προσέγγιση του Brexit θα πρέπει να είναι από τη σκοπιά των επιβατών. Ε, είναι Ευρωπαίοι πολίτες που δουλεύουν πολύ σκληρά. Το Heathrow είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο. Είμαστε βάση ε, της BA και της ε, LOT, TAP, TARON και Aegean και China αυτά και Καρούντα από την Ινδονησία. 7 εκατομμύρια, 77 εκατομμύρια συγγνώμη, επιβάτες θα έχουμε φέτος έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτες για να εργαστούν, να σπουδάσουν, για διακοπές ή ε, για να ε, μεταβούν σε άλλο τελικό προορισμό 70 με 80 ε, μακρινές αποστάσεις που δεν εξυπηρετούνται από άλλα αεροδρόμια. Είναι κόμβος λοιπόν το Λονδίνο για τους επιβάτες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε αυτών των ε, υπηρεσιών. Και είναι και επίση ε, ένα μεγάλο λιμάνι, το λιμάνι του Λονδίνου, εκτός από αεροδρόμιο. Και αυτό αφορά τις εξαγωγές, και στις μεγάλες αποστάσεις τα αγαθά υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλής ποιότητας συχνά ταξιδεύουν μόνο αεροπορικός. Ε, Υψηλή τεχνολογίας ηλεκτρονικά, ε, άλλα στοιχεία που είναι ε, κρίσιμα για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Οικονομία, αλλά και για την κοινωνία. Άρα η αεροπλοεία δεν είναι ένα ακόμα κλάδο τη οικονομία, είναι εκείνο ο οποίο διευκολύνει όλους του υπόλοιπου κλάδου. Μια μικρή εταιρεία στο Ταλίν μπορεί να συναλλάσσεται με πελάτες στο Λονδίνο οι ξενοδόχοι ε, στην Ισπανία να δέχονται ε, εκατομμύρια ε, Βρετανών τουριστών ή κάποιος άλλος Ευρωπαίος να σπουδάζει στην Οξφόρδη. Το 1 τρίτο των αεροπορικών ταξιδιών όλων των Βρετανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς την Ισπανία. Είναι συνταξιούχοι αλλά και σκληρά εργαζόμενοι που θέλουν να χαρούν τον ήλιο και τις διακοπές τους. Ήταν από τα μεγαλύτερα Επιτέγματα στην Ευρώπη ο ενιαίος ουρανός. Ε, εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες ε, κυκλοφορούν από τον Γκτάν στο Κάσκα, από ε, άλλα σημεία στη Γλασκόβη. Αυτά τα δρομολόγια δεν θα μπορούσαν να είναι προσιτά σε τιμές που δεν θα μπορούσε κανείς να ονειρευτεί πριν από τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Αυτό είναι προς όφελος και των 27 κρατών μελών και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Μας λένε να μην περιμένουμε συμφωνία για την αεροπλοεία με τον Brexit. Τι σημαίνει αυτό. Είναι σημαντικό για το εμπόριο, αλλά δεν υπάρχει ε, συμφωνία του ΠΟΕ για να αναδιπλωθούμε όπως υπάρχει σε άλλους τομείς. Μας λένε ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στο status quo πριν το 1973, πριν πέσει το τείχος του Βερολίνου πριν εμφανιστούν οι εταιρείε χαμηλού κόστους για επιλογές και ανταγωνισμό. Άρα κάποιες ε, χώρες ε, της Ανατολικής Ευρώπης και τμήματα της Γερμανίας δεν θα έχουν πρόσβαση στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Θα υπάρχουν μικρότερες δυνατότητες διασύνδεσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα έχουμε λιγότερους ζωντανούς τουρίστες που θα ε, δαπανούν τα χρήματά τους στην Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία ή Ελλάδα. Μην αφήσετε κάτι τέτοιο να συμβεί. Θα ήταν τεράστιο σφάλμα αυτό και έλλειψη ηγετική τάση, αν δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για την αεροπλοεία, με συνέπειε άμεσε για του πολίτε που εσεί εκπροσωπείτε. Καμία συμφωνία σημαίνει ότι θα ε, έχουν ε, αποτύχει και θα απογοητεύσουν τους ε, πολίτες, ψηφοφόρους και φορολογουμένους. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους επιβάτες, αλλά και τα εμπορεύματα. Τα αεροπορικά εισιτήρια δεν προστατεύονται, τα εμπορεύματα προστατεύονται μέχρι το 2019. Γνωρίζουμε όλοι ε, ότι όταν υπάρχει ανασφάλεια, αστάθεια, δεν προσελκύεις επενδύσεις, ε, ούτε μπορείς να κάνεις προσλήψεις. Χρειαζόμαστε μια βεβαιότητα ε, δικαίου, όχι μόνο για τους αερομεταφορείς και τα αεροδρόμια, για τον τουρισμό, για τα πανεπιστήμια, για κάθε κλάδο της οικονομίας, εξαγωγή, εμπόριο. Αυτό ε, μπορεί να γίνει με ε, το να οριστεί ως προτεραιότητα η αεροπλοεία ε, στην φάση των συζητήσεων, τη δεύτερη φάση για το άρθρο 50. Για το μέλλον θα πρέπει να έχουμε εξασφαλισμένη πρόσβαση στην αγορά όσο γίνεται απρόσκοπτη και να παραμένει ε, στην ε, ενιαία αγορά της αεροπλοείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που μετράνε περισσότερο, οι πολίτες, οι επιβάτες, το συμφέρον τους θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας κατά τη διάρκεια και μετά τις διαπραγματεύσεις. Να μπορούν απρόσκοπτα να κυκλοφορούν, να εμπορεύονται, να ταξιδεύουν ε, χωρίς καμία αλλαγή. Η Επιτροπή σας μπορεί να εξασφαλίσει κάτι τέτοιο και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και να συνεργαστώ μαζί σας και με τους συναδέλφους μου προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Κάη και ευχαριστούμε γιατί μείνατε εντός του χρόνου Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κέβιν Τόλαντ που είναι επικεφαλής του αεροδρομίου του Δουβλίνου. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Με λένε Κέβι Τόλαντ, είμαι ε, διευθύνων σύμβουλος της εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο του Δουβλίνου και το Κόρκ στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία είναι με κρίσιμο τρόπο εκτεθειμένη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους τρόπους πρόσβασης, γιατί το 90% γίνεται μέσω αέρας και 78% από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το, Δουβλίνο, το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ήταν ένα από τα ταχύως αναπτυσσόμενα πέρσι στην Ευρώπη. Εξυπηρετήσαμε 23 αεροδρόμια στο Ενωμένο Βασίλειο και 30% των επιβατών που περνάνε από τράνσιτ το κάνουν μέσω ε, Δουβλίνου. Το αεροδρόμιο του Κόρκ είναι το δεύτερο αεροδρόμιο στη χώρα. Εξυπηρετούμε 13 αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου και εξαρτώμαστε κατά 58% από την κίνηση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε από τότε που ξεκίνησε το project για τους ανοιχτούς ουρανούς ότι έχει πέντε δεκαπλασιαστεί ο αριθμός των δρομολογίων με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει δεκαπλασιαστεί ε, τα δρομολόγια με ευρωπαϊκές ε, εταιρείες. 5 εκατομμύρια επιβάτες πριν από την απελευθέρωση, 28 εκατομμύρια επιβάτες περίπου πέρσι. Αυτό έχει δώσει τεράστια ωφέλη στην Ιρλανδία. Θα ήθελα να σας δείξω την επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε το, το αεροπορικό μας δίκτυο από 36 δρομολόγια σε 127 συνδέσεις, 127 δρομολόγια το 2016 για ακόμα μεγαλύτερη συνδεσιμότητα. Το Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργεί βεβαίως προβλήματα αποφασίζοντας να αποχωρήσει το 53% της κίνησης είναι μεταξύ της Ευρώπης των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Είμαστε η χώρα που εκτίθεται περισσότερο στο Brexit και η Γαλλία και η Γερμανία είναι βασικοί διαπραγματευτές και 6-7% της εναερίας κυκλοφορίας τρέφεται με τρίτες χώρες. Βλέπετε λοιπόν ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου ισότιμη σε ό,τι αφορά την αεροπλοεία. Η Ιρλανδία κινδυνεύει να έχει ανεπανόρθωτη έκθεση, ενώ οι βασικοί διαπραγματευτές όχι και τόσο τα περιφερειακά αεροδρόμια εκτίθεται περισσότερο σε αυτό το χάσμα και υπάρχουν υψηλά ποσοστά αεροδρομίων που εξαρτώνται από την ε, κυκλοφορία και την σύνδεση με πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε κάθε χώρα υπάρχουν τέτοιου είδους αεροδρόμια και η έκθεσή τους διαφέρει. Εδώ βλέπετε τα τελευταία 25 χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλο συσχετισμός μεταξύ των τάσεων για το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αεροπορικές μεταφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κανείς δεν λέει ότι θα βελτιωθεί μετά τον Brexit η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι τάσεις είναι πολύ αρνητικές. 42% των τουριστών έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και 44% των επιχειρηματικών ταξιδιών γίνονται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τουρισμό είναι βασικό για τα αεροδρόμια μα. Μιλούμε για ένα δις ευρώ ε, βιομηχανία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Ένα στους εννιά ε, ε, εξαρτάται από αυτό. Η Ιρλανδία ανταγωνίζεται τη Σκοτία, την Ουαλία, το Τέβον και άλλα μέρη και νομίζουμε ότι θα πληγούμε ιδιαίτερος καθώς ο χρόνο προχωρούν διαπραγματεύσεις για το Brexit. Το 75 με 80% της κίνησης έχει να κάνει με ψυχαγωγή από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα ε, πληγεί επίσης. Εδώ να σας πω ότι όλα αυτά τα πολλοί λένε ότι τα φανταζόμαστε, ότι είναι η κορυφή του παραγόμου, ότι δεν θα συμβούν. Όμως εμείς ε, ε, η κίνηση στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου έχει αυξηθεί κατά 6% Έχουμε πολύ καλές επιδόσεις ε, πτήσεις από την Ιρλανδία, αλλά και ε, η συνεργασία με την Βόρειο Αμερική, τη Μέση Ανατολή είναι απρόσκοπτη. Βλέπουμε δηλαδή ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Τώρα, βασικές δράσεις. Είναι βασική η πρόκληση να διατηρήσουμε τη συνδεσιμότητα με ε, τη ΣΥΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που αυτές οι χώρες υιοθετούν μια πιο ε, επιφυλακτική στάση. Θέλουμε να παραμείνουμε συνδεδεμένοι ως νησί, ε, συνδεδεμένοι και με την, το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, αλλά και με την ε, υπόλοιπη Ευρώπη και θέλουμε να έχουμε ένα παράλληλο διάδρομο στο Δουβλίνο και θέλουμε ο ενιαίος ουρανός να παραμείνει ο Μάρτιος του 2019 φαίνεται να είναι πολύ μακρινός, δεν είναι όμως καθόλου και πρέπει όλοι να ξέρουμε τι είναι ο καθένας έτοιμος να παραχωρήσει, τι είναι ο καθένας έτοιμος να ψηφίσει. Τώρα, τουρισμό ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Στον κοινό ταξιδιωτικό χώρο πρέπει όλα να διατηρηθούν. Έχουμε κοινέ ρυθμίσει για το καθεστώ των θεωρήσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να διατηρηθεί. Η Ιρλανδία είναι βασικό παίκτη και συμμετέχων σε αυτό το ζήτημα και δεν θα πρέπει να έρθει σε μειονεκτική θέση λόγω των δράσεων που αναλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει να ε, κατοχυρωθούν και να αναγνωριστούν οι ρυθμίσει σαν για την Ιρλανδία. Έχουμε ασφάλεια και κοινά πρότυπα και δεν χρειαζόμαστε διαφορετικές ρυθμίσεις. Και τέλος, κατά πόσο θα υπάρξουν επιχειρηματικέ ευκαιρίες. Ναι, θα επανεγκατασταθούν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίε που εδράζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλού και αυτό θα είναι σημαντικό για εμάς ή θα επιστρέψουν τα δασμολόγητα ε, προϊόντα για τις ε, πτήσεις προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως θα αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις ευκαιρίες. Συνοπτικά λοιπόν, ανησυχούμε ιδιαίτερως, ο κίνδυνος είναι πραγματικός από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε οι πιο εκτεθειμένοι. Πρέπει να επιληθεί το ζήτημα γρήγορα και με μεγάλη σαφήνεια για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τόλαντ, να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Golden που είναι ένας από τους εκπροσώπους των αεροδρομίων ε, του Παρισιού, των Παρισίων. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες της Προέδρου, θα προσαρμόσω την εισήγησή μου, ώστε να μην επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι από τα άλλα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια των Παρισίων είναι επίσης ε, μέλη της, μέλος της και θα θέλαμε θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτά τα λεπτά που έχω διάθεσή μου για να σας ξαναπώ ότι από την εμπειρία που ζήσαμε μετά από 25 χρόνια μιας ενίας αγοράς που έχει μεταμορφώσει σε τεράστιο βαθμό τις αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη θα σας κάνω μια χρονολογική αναδρομή. Η Ευρώπη, χάρη στην ενιαία αγορά, έχει ζήσει με πιο δομημένο και λιγότερο επαναστατικό τρόπο και δραστικό τρόπο τις αλλαγές αυτές. Μια ενιαία αγορά, μια απορρίθμιση που άρχισε ιστορικά στις ΗΠΑ και που ωφέλησε την Ευρώπη από την εμπειρία της βέβαια, αλλά με τα πλονεκτήματα που μας προσεφέρει η Ευρώπη, δηλαδή μια σταδιακή άνοδο, ε, ολοκλήρωση της ενίας αγοράς και των κανόνων που διέπουν την αεροπλοεία, τις αεροπορικές μεταφορές και έτσι σιγά σιγά προχωρήσαμε στη σημερινή, φτάσαμε μάλλον στη σημερινή κατάσταση. Αυτή είναι η αγορά. Έχει τελικά, είχε τελικά ως αποτέλεσμα και ως επιτυχία πολύ θετικό αντίκτυπο στις οικονομίες μας, στις, την οικονομία των αεροπορικών μεταφορών, της άλλαξε ε, κάθετα και το αεροδρόμιο Charles de Gaulle μπορεί να είναι ένα παράδειγμα γι' αυτό, γιατί σήμερα εκεί και λειτουργεί το hub της Air France και της KLM αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην ενιαγωρά και χάρη στις διάφορες εξελίξεις αυτής που όμως έχει και την EasyJet που μαζί με άλλες εταιρείες που βρίσκονται σήμερα εδώ, εκπροσωπεύονται εδώ, χαίρει των οφελών αυτής της ενιαίας αγοράς. Αν δούμε λοιπόν τι συνέβη στη διάρκεια αυτών των τελευταίων 25 χρόνων, η ενιαία αγορά επέτρεψε τη σύναψη συμμαχιών μεταξύ αεροπορικών εταιριών αλλά και αεροδρομίων ώστε να αναπτυχθεί διαρκώς η ε, αεροπλοείας προς όφελος πιανού, προς όφελος των επιβατών, των πελατών, οι οποίοι μπόρεσαν ταυτόχρονα να ε, χρησιμοποιούν αεροπορικές μεταφορές που τους, επέτρεψε, του επέτρεψαν να ανοιχτεί σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επέτρεψε επίσης τον Ευρωπαίο πελάτη να χέρι αεροπορικών μεταφορών που έχουν εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχουν δώσει πρόσβαση ε, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Και αυτή η νέα αγορά επέτρεψε ταυτόχρονα να ανοίξει η Ευρώπη προς τον κόσμο, να ανοίξει ο κόσμος προς την Ευρώπη, αλλά και να δοθεί η όρεξη την, ε, στους ε, Ευρωπαίους να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το μεγάλο όφελος θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ε, να έχουμε αυτό το νόημα στο μυαλό μας στις διαπραγματεύσεις. Για τους Αλδεγκόλ 30% των ε, πιβατών είναι σε, σε transfer ε, και έτσι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των διεθνών προορισμών. Και πάλι αυτό είναι αποτέλεσμα της ενιαίας αγοράς. Τα ωφέλη υπάρχουν και για τα μεγάλα αεροδρόμια αλλά και για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Στη Γαλλία έχουμε αρκετά αεροδρόμια που έχουν ωφεληθεί από την ενιαία αγορά με γραμμές που άνοιξαν παντού στην Ευρώπη από εταιρείε που δεν είναι καν ε, χώριε αναγκαστικά εθνικέ, ε, αλλά που επιτρέπουν ε, να ανοίξουν αυτά τα επαρχιακά αεροδρόμια προς διάφορες πρωτεύουσε ή ευρωπαϊκούς προορισμούς. Αυτό λοιπόν ωφελεί του επιβάτε, αλλά και την απασχόληση και όλου όσοι απασχολούνται σε ένα αεροδρόμιο και αυτούς που ζουν από τη δραστηριότητα που γεννά το αεροδρόμιο τουρισμός βεβαίως, αλλά και διάφορες ε, δραστηριότητες σχετικές ε, που δεν είναι δευτερεύουσες, αλλά δραστηριότητες ε, υλικοτεχνικής υποδομής, μεταφοράς φορτίων και ούτω καθεξής. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτήν την ιστορική αναδρομή για να δούμε πού έχουμε φτάσει, το βασικό μου μήνυμα για το μέλλον και για τις συνέπειε του Brexit είναι να πω ότι μαζί με την Ευρώπη φτάσαμε και οικοδομήσαμε αυτήν την ε, σημερινή Ευρώπη Ωστόσο, τώρα αντιμετωπίζουμε αβεβαιότητα. Είμαστε σε μια φάση αβεβαιότητα και οι αεροπορικέ μεταφορέ δεν συμπαθούν την αβεβαιότητα. Χρειάζεται ο τομέα μα αρκετού κανόνε να... και εκ των προτέρων του γνωρίζει για να μπορεί να λειτουργήσει. Δεν συμπαθεί τι απότομε ρήξει. Αυτό και είπαμε και στους διάφορους αρμόδιους που θα διαπραγματευτούν το Brexit να προσπαθήσουν να φτιάξουν κανόνες όσο γίνεται πιο γρήγορα και όσο γίνεται πιο απλώς. γιατί ο χρόνος των αεροπορικών μεταφορών και των αεροπορικών εταιριών είναι απαραίτητος ο χρόνος για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες και είναι μια πρόκληση που θα έχουμε μπροστά μας για να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Είναι ένας κόσμος που χρειάζεται κάποιους μήνες ή ίσως και ένα χρόνο για να προσαρμοστεί σε αυτούς τους νέους κανόνες που μπορεί να αποφασιστούν λόγω του Brexit. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που με ακούσατε. Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ ε, για τις εισηγήσεις σας αυτές. Θα δώσουμε αμέσω το λόγο στους συντονιστές των ομάδων μας ε, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα στον καθένα. Ναι, κύριε Βοντεκάμπα, περιορισμένο χρόνο θα σας δώσω. Θα έχετε ο καθένας τρία λεπτά για να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Και στη συνέχεια, ανά πολιτική ομάδα, θα ακούσουμε ένα άνθρωπο, ένα άτομο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ολλανδικά για κάνω και προάθηση και διαφήμιση της γλώσσας. Μισό λεπτό κύριε Βαντανκάμπ. Εντάξει με τα ακουστικά έχετε βρει όλη τη γλώσσα σας, παρακαλώ. Είναι μεγάλη τιμή μου να μιλώ με τον κύριο Χόλαντ, μια που είμαι και Ολλανδός. Έχω συγκινηθεί. Η πρώτη μου ερώτηση είναι προς τον κύριο Χόλαντ. Πώς βλέπετε το μέλλον ε, για το κοινοτικό και εκτιμένο. Τώρα έχουμε πάρα πολλούς κανόνες στην Ευρώπη που ε, βρίσκουν άμεση εφαρμογή στο Heathrow. Πόσα θα κρατήσετε από αυτά, τι θέλετε να κάνετε, θα κάνετε ένα επιλεκτικό ε, shopping και πώς το, πώς το προσεγγίζετε. Κρατάμε κάποιους και άλλους, όχι. Μετά, μια ερώτηση και προς τον κύριο Χόλαντ και προς τον κύριο Τόραντ. Μα τι ονόματα είναι αυτά, Χόλαντ και Τόραντ, δυσκολεύομαι. γιατί είναι άσα; Έχει κάποιους κανόνες που ισχύουν και στα αεροδρόμια και στο μέλλον τι θα κάνετε. Οι Βρετανικοί αερολιμένες θα εξακολουθούν να πληρούν τα ίδια κριτήρια και μπορείτε να μας πείτε κι εσείς κάτι για το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ε, εκτός, μετά το πολιτικό Brexit, έχουμε και ένα πρακτικό Brexit. Ε, όπου θέλουμε να διατηρήσουμε πολλά από τα κεκτημένα. Εγώ δεν θέλω καθόλου να γίνει πόλεμος. Ας διατηρήσουμε την ανοιχτή ε, εικόνα και φιλελεύθερη των αερομεταφορών. Αυτά τις ερωτήσεις είχα, γιατί με... Ε, μου δώσετε το λόγο πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζα. Ε, σοσιαλιστές, ποιος θέλει το λόγο. Ο κύριος Λιμπεράτσκι, παρακαλώ. So following I'll be promoting Και εγώ, ακολουθώντας τις τάσεις, θα προωθήσω την πολωνική γλώσσα και θα μιλήσω στα πολωνικά. Είμαι εντυπωσιασμένο κυρίε και κύριοι, με τα πολύ θετικά λόγια που είχατε να εκφράσετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καιρό είχαμε να ακούσουμε τόσα καλά πράγματα για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, οφείλω επίσης να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένο διότι έχετε συνειδητοποιήσει πλήρως πόσο τεράστιες θα είναι οι συνέπειες του Brexit. Και στρέφομαι προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του αεροδρομίου του Χήθρο για να μας πει αν ψήφισε υπέρ της αποχώρησης ή υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν άκουσα όμως τίποτα για ένα σχέδιο Β. Τι θα γίνει εάν υπάρξει τελικά σκληρό Brexit και οδυνηρό. Πώς θα λειτουργήσουν τα αεροδρόμια, πώς θα συμπεριφερθούν, πώς θα αντιδράσετε. Γιατί έχουμε μια ιδέα για τις ε, συνέπειες και για τη βλάβη και γι' αυτό απευθύνεται και έκκληση για τη διατήρηση του συστήματος των ενιαίων ουρανών. Όμως δεν είπατε λέξη για το τι θα συμβεί εάν υπάρξει σκληρό Brexit. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ευχαριστώ. Ο προ... Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Ζήλε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Η παρέμβασή τους ήταν ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης. Δεν θα καθίσω πολύ, πρέπει να προλάβω την πτήση μου και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό και, γι αυτό και σας εξηγώ το λόγο. Όμως, ας φανταστούμε ότι ο κύριος Μπαρνιέ δεν θα έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική εντολή από αυτή που έχει τώρα του χρόνου το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2018. Με αυτό το δεδομένο, τι περιμένετε να συμβεί στην επιχείρησή σας, στην επιχειρηματική δραστηριότητα των αεροδρομίων. Μέχρι σήμερα ο κύριος Μπαρνιέ είπε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία για τα χρηματοπιστωτικά και για τα δικαιώματα των πολιτών, δεν θα υπάρχει συμφωνία και για τα υπόλοιπα και δεν θα υπάρξει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Έχουμε και τον κοινό ευρωπαϊκό ε, χώρο αεροπορίας και το Κοινοβούλιο κάνει το κομμάτι που του αναλογεί. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εκπληρώνει όλο το κοινοτικό και εκτιμένο για το θέμα αυτό. Η Βρετανική πλευρά θέλει κάποια πράγματα να τα βγάλει εκτός και εκτιμένου ή θέλετε να γίνει πλήρη επαναρρύθμιση και να μην πληρώσετε για την πρόσβαση για τον ενίο χώρο όπως δεν θέλετε να πληρώσετε για τις χώρες της Βαλκανικής, οι όπως και οι χώρες Βαλκανικής οι οποίες ανήκουν στον ε- κοινό ευρωπαϊκό εναέριο χώρο χωρίς να είναι χώρες μέλη όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ τον κύριο Ζήλε για το Άλντε, για τους φελελεύθερους. Η κυρία Μπιλμπάου. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους παρεμβαίνοντες γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπαν. Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα στον κύριο Τζον Χόλαντ. Πώς αντιμετωπίζετε όλους αυτούς τους μήνες που έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για το Brexit, τα θέματα αυτά. Έχετε νούμερα αριθμητικά, έχετε στοιχεία, έχετε δεδομένα που να δείχνουν ότι υπάρχει άμεσος αντίκτυπος ε, λόγω αυτής της απόφασης ή νούμερα που να δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή πάρτε ενδεχομένως καλύτερα. Ή, τα στοιχεία δείχνουν ότι περιμένετε τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης. Θα θέλαμε να ξέρουμε δηλαδή ποιο ήταν, ε, πώς επηρέασε το δημοψήφισμα. Από εκεί και πέρα. Υιοθετείτε κάποιο μέτρο εν ώψη ενδεχομένης αποχώρησης που δεν ξέρουμε ποια μορφή θα λάβει. Και νομίζω ότι όλοι οι βουλευτέ πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Ψηφίζουμε κάποιε γενικέ γραμμέ στη διαπραγμάτευση και σε αυτό το πρώτο γύρο διαπραγμάτευση στι 19 Ιουνίου καθορίστηκαν οι προτεραιότητε, δηλαδή το καθεστώ των Ευρωπαίων πολιτών και Κατά δεύτερο λόγο, το τιμολόγιο, η τιμή, ο λογαριασμός που θα πρέπει να πληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο πριν αποχωρήσει. Αυτό είναι κάτι που κάνουν ε, αποδεκτό όλα τα θεσμικά όργανα και όλοι οι βουλευτές. Και τέλος, σε σχέση με την Ιρλανδία, έχουν ακουστεί κάποιες φωνές ε, μέσα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ότι δηλαδή, εάν κάποια στιγμή η Βόρειος Ιρλανδία αποφάσιζε να συγχωνευτεί με την Νότιο, τότε η απόφαση θα είναι αυτόματη. Αξιολογήσατε αυτή τη δυνατότητα, ποια ο αντίκτυπο θα έχει στην πραγματικότητα των αεροδρομίων, ε, στα οποία αναφερθήκατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταλούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αξιοποιήσω την ευκαιρία και να μιλήσω τη μητρική μου, τη Σουηδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους προσκεκλημένους. Οι συνέπειες του Brexit θα πρέπει να περιοριστούν όσο γίνεται περισσότερο. Και σας ευχαριστώ που το είπατε. Εμείς οι πράσινοι αγωνιζόμαστε έτσι ώστε να αποτραπούν αυθαίρετες αρνητικές συνέπειες στην γεννητικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων ή όσο γίνεται να περιοριστούν. Γιατί δεν θα πρέπει να είναι το Brexit εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα συζητούμε τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, τα ενεργειακά και δεν θα πρέπει να περιορίζεται, επαναλαμβάνω, η κυκλοφορία των Ευρωπαίων. Τι μπορούν να κάνουν οι Ιρλανδοί, γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της Ιρλανδίας προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ, κυρία Γιούτο. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν κατά το εσωτερικό των μελετών, των αναλύσεων για τις ενδεχόμενες, ε, τον, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των μεγάλων hub στην Ευρώπη, λαμβάνεται υπόψη τη, ε, τον αντίκτυπο που θα έχει το Brexit στα μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία του, της κυκλοφορίας αυτά τα αεροδρόμια ε, που, διατηρούν, ε, που διατηρεί δηλαδή ζωντανά αυτά τα αεροδρόμια ε, είναι αυτές οι low cost εταιρείε. <clears throat> Ακριβώς επειδή μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε κράτος μέλος όπου είναι διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχουν την έδρα τους και έτσι λοιπόν έχουν ε, πάρει ζωή, πάρει ανάσα αυτά τα μεγάλα, τα μικρά μάλλον περιφερειακά αεροδρόμια. Ε, με το Brexit λοιπόν τι θα γίνει, φαντάζομαι θα το έχετε λάβει υπόψη, τι είδους ε, προσωμιώσεις έχετε κάνει για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Ευχαριστώ πολύ και τώρα για ένα λεπτό θα δώσω το λόγο σε έναν εκπρόσωπο κάθε πολιτικής ομάδας. Ο κύριος Μάρκος Πίπερ έχει το λόγο. Υπάρχουν διάφορες μελέτες και τις βολή των κοινοτήτων. Μία που λέει όλα καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα παραμείνει στην ΑΖΑ, ε, Eurocontrol, στον νέο ευρωπαϊκό χώρο, Single Europe Skype και δεν θα υπάρξει πρόβλημα με το Brexit. Εγώ όμως πιστεύω ότι όταν κάνεις το πρώτο βήμα πρέπει να κάνεις και το δεύτερο. Έχουμε το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Κάτι θα αλλάξει και θέλω να ρωτήσω τους αερολιμένες. Πού θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η αλλαγή. Έχετε κανένα προσανατολισμό. Ε, τι κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες χώρες, την Ελβετία, τον Καναδά. Εγώ δεν είμαι τώρα ο εμπειρογνώμων για να μπορώ να το κρίνω αυτό και να το αξιολογήσω. Ε, υπάρχει ένας προσανατολισμός για το προς τα πού θα αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Κύριε Πίπερ, σοσιαλιστές, ποιος θέλει να κάνει ερώτηση. Η κυρία Λούση Άντερσον. Κάτι άλλο ήθελα να πω αργότερα για τους κατασκευαστές και την αεροδιαστημική ε, ε, βιομηχανία. Τώρα για το Brexit. Είναι σαφέστατο ότι το να μην υπάρχει καθόλου συμφωνία δεν είναι σε καμία περίπτωση καλύτερο από κάποια συμφωνία. Και αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας. Όλοι είμαστε περήφανοι Ευρωπαίοι. Ό,τι και να γίνει, δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια μαζική ανασφάλεια και βεβαιότητα και χαίρομαι που το αναφέρετε κι εσείς αυτό. Να ρωτήσω όμως, ποια είναι η άποψή σας για τους εργαζομένους και την απορρίθμιση. Θα αναφερθούν και επόμενοι ομιλητές σε αυτό. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να προκύψει μια κατάσταση όπου οι εργαζόμενοι ανά την Ευρώπη ε, εξωθούνται προς τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή και τα ε, δικαιώματά τους, η προστασία των εργαζομένων δεν είναι δεδομένη και σεβαστή. Επίσης, στην ε, εφοδιαστική αλυσίδα, μία ερώτηση. Α, εντάξει, ένα ακόμα. Σε όλα τα κρατη της Ένωσης, Υπάρχουν εξαρτήματα, αγαθά, υπηρεσίες που εξακολουθούν να κυκλοφορούν. Πώς θα γίνει αυτό στα πλαίσια ε, της γενικής ανασφάλειας που βλέπουμε να επικρατεί στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Κυρία Φώστερ. Thank you very much and Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για τις παρουσιάσεις. Έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Καταρχάς για αυτά που είπε ο Τζον για το Χήθρο. Είπατε ότι θα επιστρέψετε στο 1973. Εγώ ήμουν υπέρ της απελευθέρωσης της ε, βιομηχανίας αυτής στη δεκαετία του 80. Πιστεύετε ότι πράγματι χρειάζεται να πάμε τόσο πίσω. Εγώ νομίζω όπως όχι. Και για το Δουβλίνο μιλήσατε για τα πρότυπα ασφαλείας. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, θα ε, συμμορφωθούμε σε θέματα ασφαλείας. Είναι όλα τα μέλη της ICAP. Θα παραμείνει καταστατική νομοθεσία στον Ενωμένο Βασίλειο. Περιμένω να υπάρχει αρκετή μεταβατική περίοδος εάν χρειαστούν αλλαγές ούτως ή άλλως. Και ως προς τη συμμόρφωση Πώς ε, δεν θα σα ολοκληρώσει και δεν θα εκπληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο το κεκτημένο. Εγώ δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαν Μίλτεμπεργκ. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα για την ε, ΕΑΣΑ στον κύριο Κάι. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μέλος της ΕΑΣΑ, ποιες θα είναι οι συνέπειες. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε και για τις αρμοδεότητες της ΕΑΣΑ. Για εξοπλισμό που σχετίζεται με την ασφάλεια και διάφορα θέματα. Ποια είναι η θέση σας. Είστε υπέρ του να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο μέλος της ΕΑΣΑ. Ε, προβάλλετε τέτοια επιχειρηματολογία εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσπαθείτε να επηρεάσετε την διαπραγματευτική θέση. Τώρα είστε μέρος ενός ατελούς ευρωπαϊκού εναέριου ουρανού, εναέριου χώρου. Είστε μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών TNT. Θα θέλετε να παραμείνετε σε αυτά και σε πρωτοβουλίες όπως ο Κέσαρας, το Σεζάρ. Ευχαριστώ, κύριο Κράμε. Ε, δεν θα υπάρξει επιλεκτική ε, προσέγγιση. Έχουμε συμφωνίες και με την Ορβηγία και με την Ελβετία, αλλά ορισμένοι πληρώνουν και αφήνουν να ακολουθούν τους νόμους. Για τους περιφερειακούς αερολιμένες, σε 10 χρόνια τουλάχιστον, πρέπει να είναι κερδοφόρα. Τα μισά περιφερειακά αεροδρόμια είναι ελληματικά. Εσείς δεν το κάνετε αυτό. Βεβαίω είναι σημαντικέ θέσει εργασία. Ποιο θα πληρώνει αυτά φορολογούμενο. Δέχεστε τελικά να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όταν φτάσουμε σε δίκες, όταν παραβιάζονται κοινωνικά δικαιώματα και άλλα. Αυτό το δέχεστε ή λέτε ότι όχι όλα θα ρυθμίζονται στη Βρετανία. Και γιατί γίνεται τώρα η συζήτηση μετά το δημοψήφισμα. Κανονικά τα αρνητικά ε, της εξόδου θα έπρεπε να τα είχατε συζητήσει εκ των προτέρων και μήπως θα έχει διαφορετική έκφαση το δημοψήφισμα. Αλλά 30 χρόνια όταν αμαυρώνεις και κατηγορείς την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά μην έρχεσαι και απορείς γιατί ο κόσμος την καταψηφίζει. Ευχαριστώ κύριε Κράμα. Η ευθυντή άλλος. Όχι. Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις έγιναν ε, στους ομιλητές μας και τι θα πρέπει να ε, κρατήσουμε ως κεκτημένο και τι κάνει ο Οργανισμός Ασφάλειας στην Αεροπλοεία, η ΆΣΑ. Επίσης, τι γίνεται με τους ε, περιφερειακούς αερολιμένες, πώς θα επηρεαστούν και αν είναι σκληρό το Brexit υπάρχει σχέδιο Β για τις υποδομές των αεροδρομίων. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά, έχουμε εναλλακτική πρόταση. τα έχετε προβλέψει. Γίνεται λόγος για την κινητικότητα και την εύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων. Μήπως χρειάζεται αύριο ένας ευρωπαϊκός συντονισμός, ρύθμιση, νομοθεσία. Για όλα αυτά θα σας δώσω το λόγο τρία λεπτά στον καθένα να απαντήσετε. Γιατί τίθενται όντως αυτά τα ερωτήματα, αλλά εσείς που είστε και πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση τα έχετε σκεφτεί. Monsieur Hollande, c'est à vous. Κύριε Χόλαντ, έχετε το λόγο. Uh, so, just for the record, I did actually campaign for the Remain vote. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν υπέρ του να παραμείνουμε στη διάρκεια της εθνικής εκστρατείας και το βασικό μου επιχείρημα ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, επιτυχία για τον φυσιολογικό άνθρωπο, τον απλό άνθρωπο, αλλά ως ήθιστε στο σπίτι μου κανείς δεν με άκουσε. Ε, τώρα όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με βάση την ισχύουσα κατάσταση. Ο η αγορά της ε, αεροπλοεία είναι ολοκληρωμένη. Χρειάζεται να έχουμε κοινά στάνταρ, κοινού τρόπου εργασία, γιατί αυτό μειώνει το κόστος, μειώνει την το περίπλοκο χαρακτήρα, είναι πολύ πιο ασφαλές. Και όσον αφορά την ΕΑΣΑ, εμείς αναμένουμε ότι θα μείνουμε μέλη της ΕΑΣΑ. Αυτό ε, θέλουμε στο, και ζητάμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίση για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και το Σέζαρ. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους πρωτοπόρους σε αυτό το σχέδιο και στο Χήθρο πιστεύω ότι είμαστε από αυτούς που νωρίτερα υιοθετήσαμε το ICDM που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το ΣΕΖΑΡ αλλά και έχουμε και ένα σωρό τεχνικές που είναι σύμμορφες. Θέλουμε να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε. Τώρα, μέχρι στιγμής είδαμε το ψηλότερο επίπεδο πεπιβατών και φορτίων εδώ και μια δεκαετία τους περασμένους 6 με 9 μήνες. Πολλά από αυτά συνδέονται με τις ισοτιμίες, αλλά νομίζω και μια αίσθηση στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι ο κόσμος απλά συνεχίζει να ζει και εμπιστεύεται εμά ότι εμείς θα κάνουμε τις καλύτερες δυνατές μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις. Το Brexit είναι πολιτικό θέμα και όχι επιχειρηματικό θέμα. Εάν αγνοήσουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των απλών εργαζόμενων ανθρώπων, τότε τα εμπορικά θέματα θα καταστούν πολιτικά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις για απασχόληση καθώς και ανάπτυξη. Και ότι θα διατηρήσουμε τα πράγματα όσο γίνεται πιο κοντά στο status quo. Νομίζω πως αυτό είναι προς το συμφέρον τόσο των Ευρωπαίων όσο και των Βρετανών τουλάχιστον όσον αφορά την αεροπλοεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Όλαντ. Ο κύριος Τόλαντ τώρα. Uh, ευχαριστώ. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Sorry if I address first. Συγγνώμη. Για την ΕΑΣΑ και ε, το ΙΚΑΤ δεν ξέρω ε, υποθέτω ότι θα πρέπει να παραμείνει αμοιβαιότητα. Δεν ξέρουμε πώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα το αντιμετωπίσει αυτό μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων. Για το σχέδιο Β δεν υπάρχει. Ο καθένας εκπονεί τα δικά του σενάρια και εμείς φυσικά ανησυχούμε πάρα πολύ. Είναι βασική προτεραιότητα ε, λόγω της εξάρτησης της Ιρλανδίας από τις συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν έχουμε ιδέα τι θα κάνουν και πώς θα ε, έχουν θα μας πούν οι επιβάτες και οι πελάτες των αερομεταφορέων, αλλά είναι παρατεταμένη η ανασφάλεια μέχρι το Μάρτιο του 2019. Για τα περιφερειακά, όπως είπε ο, ο κ. Κράμερ, ότι τα μισά περιφερειακά αεροδρόμια ε, είναι ελληματικά. Σας έδειξα προηγουμένως στο διάγραμμα πώς εκτεθειμένα είναι τα περιφερειακά αεροδρόμια. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί ο φορολογούμενος να το επομιστεί αυτό το κόστος, ούτε οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αγορά ε, που ε, επέτρεψε στις εταιρείες να μπορούν να πετάνε και στα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια και να υπάρχει ο ενίος ουρανός. Κάποιος ρώτησε για τη Βόρεια Ιρλανδία. Εγώ δεν θα τολμούσα να μπω σε τόσο περίπλοκη ε, κατάσταση. Το Δουβλίνο εξυπηρετεί όμως όλη την Ελλάδα. Δύο στους τρεις επιβάτες από όλη την Ελλάδα περνούν από το Δουβλίνο. Και ακριβώς είμαστε πιο εκτεθειμένοι. Ε, ε, και λόγω των συνόρων και λόγω της κοινή επικράτεια που κυκλοφορούν, οι τουρίστε, οι εργαζόμενοι. Αν υπάρχει ε, χάο για την η δημοκρατία της Ιρλανδίας θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το χάος για τη Βόρεια Ιρλανδία. Είδατε προηγουμένως ένα παγόβουνο. Και ε, τώρα αρχίζει η πραγματικότητα του Brexit. Ε, ε υπάρχει μια μεγάλη ανασφάλεια στο χείλος του κρεμού. Νομίζω ε, από το Δουβλίνο έχουμε 23 πτήσεις. Ε, σε βρετανικά αεροδρόμια από το Δουβλίνο, 8-9 τη μέρα για το Λονδίνο. Και αυτό είναι θέμα και διαπραγματευτική θέση και πίεσης. Ευχαριστώ κύριε Τολάντ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Νάντελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αερολιμένες που θα παραμείνουν στην ενιαία αγορά είναι εκείνοι τελικά που θα έχουν τις περισσότερες ευκαιρίες και την περισσότερη τύχη, γιατί οι επιπτώσεις του Brexit έχουν να κάνουν με τις αερομεταφορίες που δουλεύουν στα βρετανικά αεροδρόμια από και προς και θα έχουν να υποστούν τους νέους κανόνες όσοι λειτουργούν με βρετανικές άδειε. Και σήμερα ε, λειτουργούν με τους όρους ενιαίας αγοράς και αυτό μπορεί να έχει στη συνέχεια επιπτώσεις στα υπόλοιπα αεροδρόμια που θα παραμείνουν στον ευρωπαϊκό ενιαίο χώρο. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον να δούμε την έκβαση των ε, διαπραγματεύσεων. Συμμερίζομαι ε, τον προβληματισμό και τις ερωτήσεις ε, των ευρωβουλευτών. Τα λεγόμενα περιφερειακά αεροδρόμια που ζουν πολύ από εταιρείε χαμηλού κόστους που έχουν βρετανικές άδειες και σημαία προφανώς θα υποστούν τις συνέπειες και θα αναγκαστούν να τις επομιστούν. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα που θα τεθεί αύριο στους Ευρωπαίους είναι υπάρχουν κάποια οικονομικά μοντέλα εταιριών και αεροδρομίων, θα συνεχίσουν να υπάρχουν και τελικά δημιουργήθηκε αυτή η αγορά, αυτή η διάθεση των Ευρωπαίων να ταξιδεύουν έτσι με αυτόν τον τρόπο και οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να επιθυμούν να χρησιμοποιούν αυτά τα μοντέλα και αυτές τις εταιρείες. Και επειδή η φύση απεχθάνεται το κενό, θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το κενό θα καλυφθεί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς από τις χώρες που θα παραμένουν στην εσωτερική αυτή αγορά. Ευχαριστώ πολύ τους εκπροσώπους των ε, διαφόρων αερολιμένων και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ και στρέφομαι προς εσάς που εκπροσωπείτε τις εταιρείε αερομεταφορής. Ε, με τον ίδιο τρόπο, 5 με 7 λεπτά έκαστος για να μας πείτε πραγματικά πώς βλέπετε τις μελλοντικές επιπτώσεις του Brexit. Ο κύριος Willy Walsh Διευθύνων Σύμβουλο του International Aviation Group. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Η International Airlines Group είναι προϊόν της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Έχουμε καταχωρισμένη έδρα στην Ισπανία. Είμαστε εισηγμένοι στο Ισπανικό και στο Λομβρέζικο χρηματιστήριο δικού μου από το Λονδίνο έχουμε έξι, βασικές, ε, έξι βασικά σήματα αεροπορικών μεταφορών ε, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, λειτουργούμε παγκόσμια, απασχολούμε 60.000 ανθρώπους, 100 εκατομμύρια επιβάτες μεταφέραμε και εγώ ψήφισα να παραμείνει η χώρα μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι περήφανη και καλό είναι για τα επιτεύγματα που έχει να παρουσιάσει στον τομέα της αεροπορίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει μεγάλους αγώνες για την κατοχήρηση του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης, βασικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως κλάδος δεν σας έχουμε δώσει ακόμα δωρεάν μετακίνηση και σίγουρα οι συνάδελφοι δουλεύουν σκληρά για να σας δώσουν δωρεάν μετακίνηση, αλλά σας έχουμε δώσει ε, προσβάσιμες οικονομικά αεροπορικές εταιρείες που διευκολύνουν τους ανθρώπους ε, να μετακινηθούν καλύτερα, αλλά και που μεταφέρουν αγαθά και εμπορεύματα. Δεν έχουν ωφεληθεί μόνο οι λίγοι. 900 εκατομμύρια άνθρωποι πέταξαν από και προς πέρσι. Αναμένεται να φτάσουμε στο 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους φέτος από την απελευθέρωση και την απορρίθμιση της ε, αεροπορικής βιομηχανίας το 1993. Είχαμε με καλύτερο ανταγωνισμό, περισσότερες επιλογές, χαμηλότερα ε, ναύλα. Για τα εισδιαφάνειες τι θέλετε να κάνετε, ρωτάει η Πρόεδρος, ε, μπορείτε να τις αγνοήσετε. Με ενδιαφέρει περισσότερο να ακούσουμε, αυτά που έχω να πω από Ο αριθμός των ε, διαδρομών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ανταγωνίζονται περισσότερες από δύο αεροπορικές εταιρείες από 61 το 93 έχει 650 εταιρείες σήμερα. Η βιομηχανία στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα ε, του τουρισμού και του εμπορίου 210 δις ευρώ ε, και στηρίζει 3,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη των 27, το 1% του ΑΕΤ, δυσανάλογο όφελος για το Ηνωμένο Βασίλειο 87 δις και 3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Από το 2011 η IAG έχει επενδύσει 12 δις δολάρια σε, αεροσκάφη Airbus και έχουμε τρομερή προστιθέμενη αξία ύψους 60 δις Αμερικανικών δολαρίων. Περιμένουμε να μας παραδοθούν με τα φτερά κολλημένα και τα φτερά φτιάχνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο των Ερμπάς, όπως ξέρετε δεν καλύπτει ο ΠΟΕ την αεροπορία, αποκλειόμαστε από τους κανόνες του ΠΟΕ, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, άρα όταν υπάρξει σκληρό Brexit και αν υπάρξει δεν μπορούμε να αναδιπλωθούμε στην πρώτερη κατάσταση μέσα στο ΠΟΕ. Και παρόλο που έχουν γίνει κινήσεις για περαιτέρω απελευθέρωση, οι κανόνες υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Και κατά τρίτο λόγο, κάτι που είναι σημαντικό για τους καταναλωτές, η αεροπορική βιομηχανία πωλεί τα προϊόντα μας ένα χρόνο νωρίτερα. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο οι διαπραγματευτές να εστιάσουν την προσοχή τους στην αεροπορική βιομηχανία έτσι ώστε ένα δις άνθρωποι που αναμένεται να ταξιδέψουν φέτος και του χρόνου να συνεχίσουν να κλείνουν πτήσεις με τις αεροπορικές εταιρείες έχοντας εμπιστοσύνη ότι η υπηρεσία την οποία κλείνουν και ζητούν πράγματι θα παρασχεθεί από την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία. Το σύστημα των διεθνών ε, συμφωνιών για εξυπηρέτηση για ένα αέριο χώρο ε, είναι ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπογράψουν μια συνολική συμφωνία για τι αεροπορικέ μεταφορέ, πολύ πιο ανοιχτή από αυτέ που ήδη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη ΣΥΠΑ, το Καναδά και άλλε τρίτε χώρε αναγνωρίζοντας ότι είναι βαθύτερη η σχέση μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ ΙΤΑΒ δηλαδή και Ευρώπη των 27. Θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να προχωρήσει και όλες οι αεροπορικές εταιρείες από την Ευρώπη των 27 και όλες οι αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ Βασιλείου να έχουν όλες τις ελευθερίες και να μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα μεταξύ των διαφόρων εθνικών επικρατιών. Και η συμφωνία θα πρέπει να διευκρινίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες εντός Ηνωμένων Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 27, των 27 θα πρέπει να είναι στην ιδιοκτησία οποιοδήποτε μέρους χωρίς ε, περαιτέρω ανάγκη για ρυθμίσεις ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συμφωνία για την αεροπορία όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαπραγματευτέ πρέπει να βρουν τρόπο να δώσουν τη δυνατότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει μέλο τη ΕΑΣΑ, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συμβάλει καθοριστικά στην ΕΑΣΑ. Αυτό είναι αναγνωρισμένο ευρέω στην αεροπορική βιομηχανία, η, η μεγάλη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μεγάλα ωφέλη. Πιστεύουμε ότι το 40% των απασχολούμενων που δεν ανήκουν στην ΕΑΣΑ συμβάλλουν ε, στη δουλειά τη και είναι Βρετανοί και θα πρέπει να συνεχίσουν να μπορούν να συμβάλλουν στην ΕΑΣΑ. Και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι πλήρες μέλος είτε με τη μορφή μιας από κοινού επιτροπής ή κάποια άλλη διοικητική διάρθρωση. Τώρα προς την ασφάλεια ε, την ευρύτερη δεν είναι προς το συμφέρον κανενός ούτε στον Ηνωμένο ούτε στην Ευρώπη των 27 να αποδυναμωθεί η ασφάλεια ή να μειωθεί η συνεισφορά των υπρογνωμόνων και ειδικών επί των θεμάτων ασφαλείας. Είναι σημαντικά τα διακύβευματα και οι προκλήσεις. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ακραδάτως ότι πρώτα προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αεροπορία, την αεροπλοεία και να αναγνωριστεί πόσα ωφέλη έχει δώσει αυτό ο κλάδος τους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ολύρη. Κύριος Όλιρη, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά έρχομαι. Πάντα χαίρομαι να έρχομαι στις Βρυξέλλες που περνώ αρκετό χρόνο που δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ξέρετε ποια είναι η Ryanair, πιο αγαπημένη αεροπορική εταιρεία στις ευρωπαϊκές αγορές με το χαμηλότερο ναύλο. Ε, περιμένουμε να φτάσουμε στα 130 εκατομμύρια ε, ε επιβάτες. Ε, έχουμε το χαμηλότερο ναύλο και περιφερειακά αεροδρόμια για να μειώνεται το κόστος για τους καταναλωτές που πετούν. Βλέπετε, 41 ευρώ είναι ο μέσος ναύλος και ε, συμπιέζουμε το κόστος παντού στην Ευρώπη προς τα κάτω έτσι ώστε πραγματικά ε, τα επόμενα χρόνια να παραμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Ε, πραγματικά αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Θα συμφωνήσετε μαζί μου. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα που έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Την επόμενη διαφάνεια. Κοιτάξτε εδώ που πετάμε στην Ευρώπη, εντάξει, μεθεπόμενη. Έτσι θα αυξηθούμε τα επόμενα χρόνια μέχρι 200 εκατομμύρια τα επόμενα 8 χρόνια. Εγώ είμαι Ιρλανδός, ακόμα και αν υπάρξει Brexit, εμείς θα πετάμε χαροπά σε όλη την Ευρώπη, μπορεί να μην πετάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα περιφερειακά αεροδρόμια. Θα πάρουμε εμείς πολλά αεροσκάφη από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019 και θα κατευθυνθούμε στα περιφερειακά αεροδρόμια που θα δουν να ε, αναπτύσσονται ακόμα περισσότερο και ελπίζω να έχει αδειάσει τότε το Χίθρο. Ε, υπάρχει μια πραγματική προοπτική και θα πρέπει να το σκεφτούμε. Μήνες, εβδομάδες μετά το Μάρτιο 19 δεν θα υπάρχουν πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς ε, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν παραμείνει στη θέση της και εμείνει η Βρετανική κυβέρνηση, τότε θα βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ανοίξουν τα σλότς, οι χρονοθυρίδες. Άρα δεν υπάρχει στον ΠΟΕ συμφωνία και θα πρέπει ε, να βρουν έναν τρόπο να επανέλθουν στον ελευθερό ουρανό, τον ευρωπαϊκό ή να κάνουν διμερείς ε, συμφωνίες. Αυτό δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει ε, βούληση ε, και καλή προαίρεση από πλευρά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Lufthansa και Air France ε, βλέπουν μια ανταγωνιστική δυνατότητα για να πάρουν το χώρο που αδειάζει και αυτό να είναι εις βάρος της AGZ, της Ryanair και ξέρουμε πόσο, καλά, πόσο χαίρονται οι Γερμανοί και οι Γάλλοι να στριμώχνουν τους Άγγλους, είναι καλύτεροι τους. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει συμφωνία με τη Βρετανική κυβέρνηση και όταν ρωτάμε για το Plan B, προς Θεού λένε δεν υπάρχει σχέδιο Β, υπάρχει σχέδιο Γ, δεν υπάρχει Β. Ένας από τους μεγάλους θύνοντες υπουργού είπε θα συμφωνήσουμε με το Πακιστάν τότε, ε, διμερός. Ωραία. Και έτσι ε, θα ε, αποκατασταθεί η χαμένη κυκλοφορία με την Ευρώπη. Λέει ο κλάδος πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει συμφωνία για να συνεχίσουν τα μεγάλα αεροδρόμια να υπερ ε, και να βάζουν χαράτσια. δεν θα χαλάσει και ο κόσμος αν δεν υπάρχει συμφωνία, γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018, όπου ο μέσος ε, Βρετανός ε, ψηφοφόρος ε, σκέφτεται τις διακοπές του για το 19, είτε θα πρέπει να πάει στη Σκοτία με το αυτοκίνητο και να πάρει το φέρι για την Ιρλανδία και εγώ τη λατρεύω την Ιρλανδία αλλά δεν θέλω να περνάω και όλες μου τις διακοπές ούτε οι περισσότεροι Βρετανοί. Λοιπόν, αν το δείτε σε τομεακό επίπεδο, όταν αρχίζει να καταλαβαίνει ο κόσμος την πραγματικότητα ε, ε, του Brexit, να τον στοιχιώνει το Σεπτέμβριο του 2018, τότε ε, η αεροπροϊά δεν θα περιμένει μέχρι το Μάρτιο του 2019. Αν δεν έχουμε σαφές νομικό πλαίσιο για να συνεχίσουμε να πετάμε από και προς Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο, δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία ούτε νομική βάση. Αν δεν έχουμε λοιπόν από το Σεπτέμβριο λύση, θα ακυρώνουμε πτήσεις και θα ακυρώνουμε και ε, διακοπές. Θα ενθουσιαστούν Γάλλοι και Γερμανοί γιατί αυτό θα ε, στριμώξει τις άλλες ε, εταιρείε, η IAG θα τα χάσει γιατί δεν μπορεί μια ισπανική εταιρεία να λειτουργεί από το Ηνωμένο Βασίλειο ή Βρετανική από την Ισπανία ενώ θα έπρεπε, θα έχουμε ένα μέγα χάος, ένα μπάχαλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να το λύσει. Η Βρετανία θα, θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα. Θα χαθούν θέσεις εργασία στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, στον τουρισμό, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, την Ιταλία γιατί εμείς βεβαίως αντικαθιστούμε πολλά από τα δρομολόγια προς το Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανοί, Σκανδιναβοί και Πολωνοί δεν πρόκειται να μας καλύψουν ό,τι καλύπτουν οι Βρετανοί. Και τι θα γίνει μετά, τι ότι φρύ φορολόγητα θα ρημάξουν, θα κλείσουν τα μαγαζιά, δεν θα έχουν πελάτες. Καλά, μπορεί να υπάρχει ε, ε, διατλαντική κυριοφορία. Ε, τώρα αυτά πρέπει να πηγαίνουν στο Παρίσι, ο Θεός να τους βοηθήσει, στη Φραγκφούρτη ακόμα περισσότερο. Η IAG δεν θα επιβιώσει ένα σκληρό Brexit και ίσως πείσουμε τη Βρετανική κυβέρνηση ότι η λογική έκβαση εδώ θα ήταν να αγνοήσουν το δημοψήφισμα το περσινό να παραμείνουν στην Ευρώπη σε περίπτωση που το κάνουν. Δεν χρειάζεται η Ευρώπη να αφηνιάσει. Χρειάζεται ε, μια μεταρρύθμιση που ε, ε, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 10-15 χρόνια. 30 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα το αεροδρόμιο που έχετε εδώ πέρα για να μειώσει το κόστος. Και εγώ θέλω να εξακολουθώ να υποστηρίζω την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, να έρθουν όλοι στη Ράιαν για να γλιτώσουν ένα σκασμό λεφτά. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, μην αρχίσετε τώρα τον ανταγωνισμό με τα αεροδρόμια. Εδώ είμαστε για να βρούμε κοινέ λύσεις. Και προχωράμε. Δεν το λόγο στον κύριο Κέννεντι. Είστε ένας από τους εκπροσώπους των ε, Αμερικανικών ε, ε, αεροπορικών εταιριών. Κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που με έχετε καλέσει σήμερα εδώ. Ονομάζομαι Σον Κένι, είμαι επικεφαλής της Airlines for American. Είναι η βασική εμπορική ένωση που αντιπροσωπεύει τις αεροπορικές μας εταιρείες, 90% των επιβατών και των φορτίων μετακινούμε και έχουμε την American United UPS και Atlas μεταξύ άλλων. Ε, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και την εκτίμησή μου που με καλέσατε σήμερα εδώ. Έχω εργαστεί με τα δύο σώματα το και το Κογκρέσο δηλαδή στην ε, Αμερική καθώς και ως ε, σύμβουλος στο Λευκό Οίκο υπό τον πρόεδρο Ομπάμα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίπλοκο και σπουδαίο θέμα που θα επηρεάσει την Ευρώπη, τον Ηνωμένο Βασίλειο της ήπα, καθώς ε, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί οι αεροπορικέ υπηρεσίε είναι κάτι σχετικά εύκολο να το συζητήσουμε, μάλλον γιατί όλοι μας έχουμε χρησιμοποιήσει το προϊόν και πόσο πολύ του αγγίζει. Ο πατέρας μου ήταν 27 ετών όταν πήρε πρώτη φορά αεροπλάνο την δεκαετία του 60, εγώ ήμουν 5 όταν πήρα το πρώτο μου αεροπλάνο την δεκαετία του 70 και τα παιδιά μου ε, ταξίδεψαν ε, όταν ε, ήταν μόλι μηνών κάτι που ήταν πολυτέλεια έγινε καθημερινότητα, όπως λίγο και τα κινητά τηλέφωνα. Έχουμε 377 πτήσεις από τη ΣΥΠΑ ε, στις 27 χώρες της Ένωσης καθημερινά, 76.000 επιβάτες. 20% αυτών φτάνουν στην Ένωση μέσω μιας ε, στάσης στο Heathrow. Μάλιστα, το 53% όλων μας των πτήσεων περνάνε από το χήθρο, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το χήθρο για την παγκόσμια συνδεσιμότητα. Εμείς, ε, ή μάλλον η αεροπορική γέφυρα ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ κρίσιμη πτυχή ε, το σύστημα αυτό λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και υπό το φως του συστήματος οι ιστορικά οι κυβερνήσεις έχουν αποκλείσει, έχουν αφαιρέσει τις αερομεταφορές από τις εμπορικές του συμφωνίες λόγω όλων αυτών των ε, συμφωνιών. Φέτος μάλιστα κλείνουμε 10 χρόνια από την ε, συμφωνία για τους ε, ανοιχτούς ουρανούς ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμφωνία αποτελεί τη νομική βάση για τις συμφωνίες μεταξύ αεροπορικών εταιριών, συμφωνίες ανάμεσα στη Λουφθάνσα, την Air την Καελέμ κτλ. Αυτές οι επιτήσεις είτε πάνε κατευθείαν στη ΣΥΠΑ είτε στην υπηρετική Ευρώπη Ε, και έχουν συντονισμένες ε, πτήσεις, σχέδια πτήσεων, ωράρια. Αυτό σημαίνει καλύτερο συντονισμό. Ο ανταγωνισμός δε ανάμεσα στις αεροπορικές εταιρείε. κρατάει χαμηλά τα, τα εισιτήρια, τις τιμές των εισιτήριων. Την πρώτη μέρα του Brexit Επιβάτε ε, των ΗΠΑ δεν θα μπορούν να πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο θα ισχύει και για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Το είπαν και άλλοι εδώ ότι άλλε βιομηχανίε, όπω η αυτοκινητοβιομηχανία ή η Telecom έχουν χθέσει ε, αναδίπλωση εντό του ΠΟΕ. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμα και τη απουσία συμφωνίε, όμω δεν μπορούμε παρά να πούμε ακόμα μια φορά ότι η δική μα υπηρεσία δεν είναι μέσα στον ΠΟΕ και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αν δεν υπάρχουν σαφεί κανόνε. Υπάρχουν συμφωνίε που χρονολογούνται από το 50, όπως ορισμένοι από εσάς μπορεί να θυμάστε, ήταν μια περίοδος όπου τα τηλεφώνα ήταν κολλημένα στον τοίχο, δεν υπήρχαν CD, ε, ήταν ένα επιχειρηματικό μοντέλο όπου δεν υπήρχε η στεναρή οριμότηση που έχουμε τώρα και που ο κόσμος την περιμένει πλέον. Η Συμφωνία των Ανοιχτών Ουρανών λοιπόν έχει επιτρέψει τη δημιουργία των διεπηρωτικών ε, συμφωνιών. Αυτό γιατί ε, ε, επιπλοκές θα δημιουργηθούν όσον αφορά τα εισιτήρια που πρέπει να έχουν τιμές ένα χρόνο πριν. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν ο κόσμος σίγουρα τι συμβαίνει για να μπορέσουν να κλείσουν εισιτήρια για ένα χρόνο αργότερα. Άρα δηλαδή από το 18 πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι κανόνες που θα ισχύσουν. Οι αμερικανικές αεροπορικέ εταιρείες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην καταστάση του Heathrow για τις, ε, και οι 10 πρώτες αγορέ. Ε, το Heathrow είναι οι 8 αγορέ. Για μας δηλαδή δεν είναι καν επιλογή αυτή η κατάσταση. Πού είμαστε λοιπόν οι αεροπορικά, τα αεροπορικά ταξίδια είναι πανταχού παρόντα όπως και τα κινητά τηλέφωνα. Οπότε περιμένουν ο κόσμος τα ίδια πράγματα και για τις αεροπορικές μεταφορές. Δεν θα περιμένουν διακοπή ή ρήξη μετά το Brexit. Γι' αυτό αναμένουν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβούν στις κατάλληλες νομικές ενέργειες ώστε να μην υπάρξει διακοπή. Μετά, υπάρχει η δυνατότητα μια συμφωνία ανοιχτών ουρανών ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει δρόμο δηλαδή εδώ. Και η δεύτερη επιλογή, που είναι μάλλον πιο σχετική μέσα είναι κάποια είδο συμφωνία ανάμεσα στις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι ώστε να συνεχιστεί η αγορά της αεροπλοΐας που επιτρέπει τον ανοιχτό και θα αποφύγει την, ανα, την ε, ρυθμίσεις για εμπορικές συμφωνίε. Υπάρχει σύντομο βέβαια το χρονικό διάστημα που πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις, αλλά εάν διακοπούν οι αεροπορικές υπηρεσίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ένωση, θα είναι μέγα πλήγμα για όλες τις πληγές, για όλες τις πλευρές. Οι μελλοντικές ρυθμίσεις θα έχουν στόχο τις, ε, τις, ε, τους κλάδους που θα ε, επηρεαστούν περισσότερο από τη διαδικασία και εμείς σας ζητούμε να ασχοληθείτε με την αεροπλοεία κατά προτεραιότητα. εκτιμούμε το ότι έχετε αναλάβει πρωτοπόρο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούνται από το Brexit και είμαστε ανοιχτοί να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέννεντι και τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Τόμας Κρόμπ Ορίστε. είστε του ομίλου Λουφτχάνησα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι δραματικό αυτό το γεγονός για ολόκληρη την ε, Ευρώπη. Ο κύριος Ολύρη τώρα επενήχθηκε ότι το Brexit γεννήθηκε στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Όχι και για τον όμιλο Lufthansa πρέπει να σας πω ότι θα έχει βαθιές και αρνητικές συνέπειες. Γι' αυτό θα χαιρόμαστε εάν ακυρωθεί το Brexit. Δεν είναι στο χέρι μας. Αυτό που θέλουμε είναι ε, συμμετοχή στους ε, ελεύθερους ουρανούς στη μεγάλη ενιαία αγορά που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί. 25 χρόνια κλείνουν τούτη την εβδομάδα, 25 χρόνια της εσωτερικής αγοράς της αερομεταφορές. Πριν από λίγες εβδομάδες οι Ευρωπαίοι, ε, Ευρωπαϊκές Ενώσεις Αεροδρομίων και Αερομεταφορέων στράφηκαν κατά του λαϊκισμού στην Ευρώπη και ε, δήλωσαν ότι δεν μπορεί να είναι το μέλλον της Ευρώπης αυτό 60 χρόνια μετά ε, τη ε, συνθήκη της Ρώμης. Αυτά όλα ήταν πριν τις εκλογές στη Γαλλία και την Ολλανδία. Τώρα βελτιώθηκαν κάπως τα πράγματα. Έχω την ευκαιρία να μιλώ στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να σας πω τι έγινε τις προάλλες στη Γερμανία με το G20. Επρόκειτο και για δίκαιο εμπόριο, για ελεύθερο μεν εμπόριο, αλλά κυρίως για δίκαιο εμπόριο. Και από την νομοθεσία που έχουμε δει από εδώ για τα δικαιώματα των επιβατών, σήμερα αν κοιτάξουμε λίγο πιο ανατολικά, όχι δυτικά, οι πελάτες που πετούν ε, ε, στην Κίνα ή την Ιαπωνία έχουν τα δικαιώματά τους ε, εγγυημένα και όταν επιστρέφουν. Όταν είναι ευρωπαϊκή εταιρεία, αλλά όταν δεν είναι ευρωπαϊκή, αν επιστρέφουν με την Japan Airlines, δεν ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτή που εσείς θεσπίζετε. Το ίδιο και για την, εκπομπή, την εμπορία εκπομπών ρήπων στην Ευρώπη. Βερολίνο, Φραγκφούρτη, Πεκίνο, αν πετάει η Λουφθάσα θα πρέπει να πληρώσουμε. Ε, αλλά αν πετάει η εταιρεία του Κατάρ από το Βερολίνο ε, στο Πεκίνο μέσω Ντόχας, δεν πληρώνουν ε, τέλη. Θέλουμε να έχουμε ελεύθερους ουρανούς, αλλά δικαιώματα επιβατών, ελεύθερη κυκλοφορία, ευρωπαϊκό δικαστήριο. Όλα αυτά ισχύουν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, για τους αερομεταφορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Open Sky είναι ανοιχτή αρένα για όλους, αλλά δεν έχουμε τους ίδιους κανόνες παιχνιδιού. Η νομοθεσία που θεσπίζετε εσείς θα πρέπει να ισχύει για όλους που δραστηριοποιούνται και λειτουργούν στον ευρωπαϊκό αέριο χώρο για όλες τις εταιρείες, όχι μόνο τις ευρωπαϊκές. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έχουμε γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία ε, που δεν επιτρέπεται η απεργία. Δεν έχουν το δικαίωμα της απεργίας εργαζόμενοι. Εμείς ζήσαμε 15 απεργίες στη Λουφτάνσα και μια αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης θα πρέπει να προσανατολίζεται και στις 100.000 εργαζομένους που έχουμε εμείς ως όμιλος Lufthansa στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να είμαστε εμείς μειονεκτήματα ε, για τον ίδιο μας τον εαυτό καταφέραμε να αξιοποιήσουμε την εσωτερική αγορά για να επενδύσουμε. Austrian Airlines, Air Dolomiti, ε, Brussels Airlines, ακόμα και στην Ελβετία πετάει Air Dolomiti. Αλλά παντού είναι οι ίδιοι κανόνες. Αυτό που θέλουμε είναι να παραμένουμε όλοι ενωμένοι και η Λουφθάνζα και η British Airways. Έτσι ε, γίναμε οι όμιλοι αυτοί που είμαστε. Αλλά να μην ισχύει διαφορετική νομοθεσία για άλλους. Επαναλαμβάνω για την νομοθεσία που ψηφίζετε εσείς στην Ευρωπαϊκή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν παραμείνει το Brexit, που λυπούμαστε πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν πουλήσαμε την British Midland στην British Airways, επειδή ξέραμε πώς θα βγει το Brexit. Ήταν πριν από λίγα χρόνια διαφορετική απόφαση ε, εμείς θα θέλαμε να μπορούμε να συνεχίζουμε να επενδύουμε. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ανοιχτή ουρανή, ε, νομοθεσία, ναι, αλλά με σαφές κοινοτικό εκτιμένο ε, νομολογία Στρασβούργου, Βρυξελών κτλ. Δεν θέλουμε να είμαστε δεύτερης κατηγορίας εταιρείε και αερομεταφορείς, επειδή είμαστε ευρωπαϊκοί φορείς. Ενώ άλλοι να εκμεταλλεύονται την εσωτερική αγορά και να μην πληρώνουν το ίδιο με εμάς. Αυτή είναι η σαφής άποψη του ομίλου Lufthansa. Όλοι είμαστε στην ίδια μοίρα, αλλά θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια για όλους, με τους ίδιους κανόνες παιχνιδιού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Κρόπ. Θα αντικαταστήσω για λίγο την κυρία Ντελή, την ε, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο κύριος Πασκλάινερ έχει το λόγο διευθυντής της Διεθνούς Δημόσιας Πολιτικής του, το Τμήμα Εταιρικών και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ομίλου ΤΟΥΙ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολλά έχουν υποθεί για αυτά τα θέματα. Βλέπετε τις διαφάνειες, δεν θα μακρηγορήσω. Να σας πω λίγα λόγια για τον όμιλο ΤΟΥΙ. Είμαστε η μεγαλύτερη τουριστική εταιρεία στον κόσμο, 67.000 απασχολούμενοι σε όλο τον κόσμο. Έχουμε 16 κρουαζιερόπλια, λειτουργούμε και συνεργαζόμαστε με 153 αεροπορικές εταιρείες σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρούμε ότι είμαστε απολύτως ευρωπαϊκή εταιρεία. Έχουμε 1.600-1.600 υποκαταστήματα στην Ευρώπη. Έχουμε δικά μας ξενοδοχεία και περισσότερα από 20 εκατομμύρια πελάτες από 31 αγορές που ταξιδεύουν σε 180 χώρες παγκοσμίως χρησιμοποιώντας την TUI, τον όμιλο ΤΟΥΙ. Να σας δώσω τώρα λίγα στοιχεία για τη συνολική συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 1,5-3 ευρώ συνολικά η συνεισφορά του τουρισμού στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Αν δείτε αυτή τη γραφική παράσταση, αυτά τα σχέδια, τα γραφήματα, βλέπετε ότι οι πέντε μεγαλύτεροι προορισμοί είναι η Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Και τέσσερις από τους πέντε αυτούς προορισμούς η συνεισφορά του τουρισμού στο εθνικό ΑΕΠ ξεπερνά το 10%. Στην Ελλάδα είναι για παράδειγμα 18,6% ε, η συνεισφορά του τουρισμού στο εθνικό ΑΕΠ και αυτά είναι πολύ σημαντικά νούμερα που πρέπει να έχετε υπόψη σας για να έχετε τη συνολική εικόνα της κατάστασης. Στην επόμενη διαφάνεια τώρα βλέπει κανείς και αναρωτιέται ε, ποιες είναι οι δυνατότητες, γιατί βεβαίως πάντοτε είναι πιθανολογική η συζήτηση, δεν γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα. Υπάρχει μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό μιλάμε για τις πιθανές επιπτώσεις του Brexit στον τουρισμό στην Ευρώπη των 27. 21 δις ευρώ ενδυνάμει απώλειες ως προς τις δαπάνες των τουριστών, εάν γίνει το Brexit. Αυτή είναι μια εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν δούμε πώς αναλύεται ε, στους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς, βλέπουμε για παράδειγμα ότι στη Μάλτα θα υπάρξουν απώλειες 2,4% του ΑΕΠ, του εθνικού ΑΕΠ, ε, διότι θα χάσουν τουρίστες που θα ξόδευαν στη Μάλτα λόγω του Brexit. Στην Ισπανία η απώλεια του ΑΕΠ θα είναι μισό, μισή ποσοστία ε, μονάδα σε σχέση με το ΑΕΠ. Στα αριστερά της διαφάνειας βλέπετε κάποια από τα ωφέλη που έχει φέρει ο τουρισμός, ο κλάδος του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 10% ε, συνεισφέρει στον ΑΕΠ, στο ΑΕΠ, ε, τα ταξίδια και ο τουρισμός 11,6% συνεισφέρει στην απασχόληση, 26,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί από τον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε 500 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετησίω το 40% των διεθνών αφήξεων παγκοσμίω. Φτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε πώς όλα αυτά σχετίζονται με τις ροές επιβατών από το Ηνωμένο Βασίλειο και με το Brexit. Πέντε βασικές και μεγαλύτεροι τουριστικοί προορισμοί από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Ε, και οι τουρίστες από Ηνωμένο Βασίλειο προς αυτές τις χώρες ετησίως είναι πάρα πολλοί. 13,5 εκατομμύρια Βρετανοί για παρανεπιβάτες πηγαίνουν στην Ισπανία ετησίως ή τουλάχιστον πήγαν το 2016. Να πω και κάτι για τα 2,5 εκατομμύρια Βρετανών που πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το 10% όλων των διεθνών αφήξεων του Ηνωμένου Βασιλείου ε, τα 2,5 εκατομμύρια πηγαίνουν στην Ελλάδα. Επομένως, το 2,5 εκατομμύρια Βρετανών επιβατών που πηγαίνουν στην Ελλάδα είναι το 10% όλων των διεθνών αφήξεων στη χώρα αυτή. Και αυτό πρέπει να το έχει κανείς υπόψη του. Άρα είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα, γενικότερο ζήτημα και όχι μόνο βρετανικό. Εμείς έχουμε την Thomson Airways στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουμε και πέντε αεροπορικές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Δεν είμαστε ούτε με τη μία μεριά ούτε με την άλλη. Προσπαθούμε να βλέπουμε το ζήτημα μας σφαιρικά. Ένα εκατομμύριο πτήσεις γίνονται στην, ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστοίχως από τον Βρετανό Ρεμεταφορέα και από τις πέντε ευρωπαϊκές ε, πορικές εταιρείες περίπου το ίδιο νούμερο είναι προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Brexit θα μπορούσε λοιπόν να οδηγήσει σε τέτοιου είδου συμφωνίες γνωστές. Αυτό έχει ήδη υποθεί. Έχουμε τον ε, Ευρωπαϊκό Κοινό Εναέριο Χώρο. Σίγουρα θα υπάρξει μείωση των ε, ταξιδιών μετεπιστροφής, λιγότερες επιλογές, λιγότερος ανταγωνισμός. Αυτά θα είναι δυνάμει αποτελέσματα και θα έχουμε και μείωση των τουριστικών δαπανών κατά πάσα πιθανότητα εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο του σκληρού Brexit. Και τελικά ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανωμένου του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι απώλεια 210 δις ευρώ. Αυτό είναι το πιο ακραίο σενάριο όπου θα υπάρξει πάυση των αεροπορικών μεταφορών και κάποια κομμάτια θα αντικατασταθούν από μεταφορές ιδεροδρομικές με λεωφορεία ή με φεριμπότ είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο, αλλά βλέπετε περίπου την αίσθηση του πώς διαμορφώνται τα νούμερα και τι διακυβεύεται όταν μιλούμε για τον τουρισμό και το Brexit. Εδώ κάποια βασικά μηνύματα από τη δική μας πλευρά. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ευρωπαϊκός κοινό χώρος αεροπορίας και αεροπλοείας θα πρέπει να διατηρηθεί ακριβώς χάρη ε, και λόγω του γεγονότος ότι πριν από το 1992 και πριν από την απελευθέρωση της αγοράς. Είχαμε ε, συμφωνίες αεροπορικής εξυπηρέτησης, τα ASA, Air Service Agreement, τα οποία όμως δεν αποτελούν ε, επαρκή βάση. Και είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ΆΣΑ και να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο μέλος στην ΕΑΣΑ και σημαντικό να υπάρξει ασφάλεια σχεδιασμού και νομική ασφάλεια για την θερινή περίοδο ε, του 2019 για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Παστ Λάιτνερ. Με την παρέμβασή σας κλείνει αυτή, αυτός ο κύκλος παρεμβάσεων από πλευράς της βιομηχανίας φαίνεται ότι οι αναταράξεις είναι μεγαλύτερες ε, ε, και περισσότερες στον αέρα από ότι είναι στα χερσαία μέσα μεταφοράς, τα επίγεια και υπέργεια. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συντενιστές των ομάδων, ο κύριος Βιν Βαντεκάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε επανειλημμένα έχω κάνει ε, ε, αναρτήσεις στο Twitter Brexit is impossible. Και ξέρω αυτό μπορεί να βλάψει την πολιτική μου σταδιοδρομία. Αλλά εγώ μιλώ για την πραγματικότητα. Είναι ανέφικτο το Brexit. Έχω δύο ερωτήσεις στους αερομεταφορείς. Ερώτηση πρώτη. Προς τον κύριο Κέννεντι που λίγο το υπενήχθηκε. Τι σημαίνουν οι διμερείς συμφωνίες. Ο Λύρη λέει μετά το Μάρτιο του 2018, 19 μάλλον, δεν θα προσγειώνεται κανένα αεροπλάνο. Αλλά έχουμε τις παλιές διμερείς συμφωνίες διακρατικές και αυτό είναι μια θέση αναδίπλωσης. Γιατί κάτι θα πρέπει να γίνει για να πετάνε τα αεροπλάνα. Δεύτερη ερώτηση προς τη Lufthansa και την ε, IAG. Ε, είναι διαφορετική η δική σας κατάσταση γιατί το IAG πετάει και στην Ευρωπαϊκή ε, Ήπειρο, στην Υπηρετική Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά Lufthansa εδρεύει στην Ευρώπη. Έχετε διαφορές ε, στις τιμές, προβλέψει θα είναι λιγότερο ανοιχτή και ελεύθερη αγορά, κυρίως για τη Lufthansa. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος α, η κυρία Γιάλα, Σέντερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και που θελήσατε να μας καθησυχάσετε, αλλά νομίζω πως εξ αρχής θα πρέπει να, πούμε, να μιλήσουμε για την ανάγκη να έχουμε όσο γίνεται νωρίτερα όπως ισχύει βέβαια πάντα, Όσο γίνεται λοιπόν νωρίτερα, μια σαφή οργάνωση, ε, ε, γιατί όπως είπαμε, εδώ η Ευρώπη μεν θα συζητήσει αλλά σε σχέση με το χωρισμό με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ενισχύσουμε σταθερούς κανόνες. Έπειτα, κοινωνικές πτυχές και εμείς ε, ε ακριβώ όπως γνωρίζετε και παρακολουθώ στενά το τι συμβαίνει με ε, την Αμερική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια μιας ε, συγκεκριμένης ε, και θητείας μιας κυβέρνησης σε σχέση με συγκεκριμένες χώρες όπου δημιουργούνται ανησυχίες Ανησυχούμε όμως και για το γεγονός ότι οι κλάδοι των μεταφορών όλο ένα γίνονται λιγότερο ελκυστικοί για τους νέους. Μάλιστα, μόλις διάβασα μια σχετική μελέτη που έλεγε για το ευρωπαϊκό επίπεδο ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτή την υπόθεση για τους νέους και ότι και για τους νέους υπάρχει πρόβλημα, το θέμα των πληρωμάτων δηλαδή ε, και τι θα κάνουν τα πληρώματα. Άλλο πρόβλημα είναι ο τουρισμός. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά την βίζα τουρίστες από τη Ρωσία, τουρίστες από την Κίνα. Έχουμε και αυτού να δούμε τι θα του κάνουμε. Σε ένα τέτοιο Brexit όπω μέχρι στιγμή δεν πρέπει να δρεύουμε αυταπάτε. γιατί και εγώ όπω έλεγε ο κ. Βαντερκάμπ ήλπιζα αλλά εν πάση περιπτώσει εφόσον υπάρξει ρήξη δεν θα υπάρχει ε, μία μεταχείριση, μία μάλλον ε, σχέση όπως με την Νορβηγία ή την Ελβετία. Οι Βρετανοί τουρίστε θα πρέπει να έρχονται με το διαβατήριό τους και θα μπαίνω στην ουρά μαζί με αυτούς που χρειάζονται βίζα. Ούτε αυτό θα είναι πολύ εύκολο. Έπειτα σε σχέση με την ασφάλεια. Είπατε ε, αυτό το πράγμα για τα συμπολίστε. τι έγινε, δεν μπορώ να ρωτήσω. Ναι, ναι, ένα λεπτό είχαμε πει όμως. Μπορείτε να δεν ρωτήσετε, αλλά είπαμε για ένα λεπτό ο καθένας. Το hub της TAF4 για την Ιμπέρια νομίζω πως ε, ε, δεν είναι και πολύ ωραίο για άλλες εταιρείες, να χωράει και άλλες εταιρείες. Και έπειτα, να δούμε πώς θα μπορέσουμε με διεθνείς συμφωνίες ε, να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που θα έχουμε με τον Βασίλειο και πώς θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά στην πράξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ωραίο στην πολιτική είναι ότι είσαι από αυτού του ανθρώπου που είτε βλέπουν μισογεμάτο είτε μισοάδιο αυτό το ποτήρι. Εμεί πρέπει να φροντίσουμε ώστε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Έχουμε πολλές προκλήσεις, αλλά εγώ είμαι, ε, ε, ε, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί έχουμε τα καλύτερα μυαλά στην αεροπλοεία. Και νομίζω πως είναι αρκετά απογοητευτικό, ότι ενώ υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας, επικρατεί πολύ αρνητισμός, πολύ απεσιοδοξία. Εγώ θέλω να αγγίξω κάποια από αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ για τις εισηγήσεις, πολύ διαφορετικές και πολύ ενδιαφέρουσες όλες. Συμφωνώ με τον Will Walsh που είπε ότι πρέπει να βρούμε τρόπο μέσω των συμφωνιών υπηρεσιών, συνολικές καθολικές συμφωνίες με ολόκληρο την Ευρώπη, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ομαλή μετάβαση από τη στιγμή που θα έχει γίνει το Brexit. Γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό και για τις ρεπορικές εταιρείε από τα άλλα κράτη-μέλη. Τώρα, παρά αυτό και ως, από προσωπική άποψη και ως εισηγήτρια που έχω ασχοληθεί με κάθε ε, νομοθεσία που αφορούσε την ΕΑΣΑ, τον Ενιό Ευρωπαϊκό Ουρανό, την ασφάλεια των αεροδρομίων εδώ και 17 χρόνια, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πώς έχουν εξελιχθεί όλα αυτά και γι' αυτό είμαι πολύ περίεργη και διαρωτώ με γιατί υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι μπορεί εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα θέλουμε να συμμορφωθούμε, ενώ εμείς σπρώξαμε για όλες αυτές τις αλλαγές. Αυτή είναι μια ερώτηση λοιπόν για όποιον θα ήθελε να την απαντήσει. Επίσης μιλήσατε για την ιδιοκτησία και τον έλεγχο και από τον συνάδελφο από τη είπα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε για τους ανοιχτούς ουρανούς και ήμουν εδώ και για αυτό το θέμα, ότι δεν έχουμε λύσει το θέμα του ποιος ελέγχει. Και συμφωνώ με τα όσα είπα ο για το ότι πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί υπάρχει ακόμα δυσπιστία και δισταγμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά πραγματικά, Νέα, θα μας λείψετε. Δεν θέλουμε να φύγετε από το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν πρέπει να μα το λέτε όλη την ώρα, γιατί κάποιο άλλο θα έρθει και θα σα πάρει τι δουλειέ. Και αυτό θα είναι υπέρ, υπέρ είμαστε της επιλογής για τους καταναλωτές. Εγώ ως ε, ο πρώην υπάλληλο ε, μιας αεροπορικής εταιρείας πιστεύω πάντα πως πρέπει ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει. Είναι σπουδαία η αγορά και έχουμε μεγάλες επιτυχίες. Οπότε μη φεύγεις μη Μάικλ, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε λύσεις. Ε, και πάλι νομίζω θυμόμαστε τις ημέρες όταν εγώ δούλευα για μια αεροπορική εταιρεία, ήταν η πρώτη δυτικοποιημένη ε, εθνική εταιρεία, όταν οι αμερικανικές εταιρείες ήταν ήδη στο κεφάλαιο 11 και εμείς ήμασταν ακόμα κρατικοδίαιτες εταιρείες στην Ευρώπη όλες οι αεροπορικές. Η Ατλαντική και η νησί αεροπλοεία είναι κλειδί και δεν πρέπει να υπάρξει κανένα μπλοκάρισμα εκεί ενώ συνεχίζονται αυτές οι διαπραγματεύσεις και φυσικά και όταν θα γίνει η μετάβαση. Τέλος, ο Τόμας με τη Λουφτχάνσα. Δεν θα δούμε το 8-6-8 που αφορά τον ανταγωνισμό. Αυτό θα είναι συζήτηση κάποια άλλη μέρα. Αλλά μένα με ανησυχούν ε, αυτές οι, οι πόνοι προστατευτισμού που ακούγονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από Ευρωπαίους μεταφορείς που δεν θέλουν ανταγωνισμό από τρίτες χώρες από ό,τι φαίνεται. Και επίσης προσέχετε τι εύχεστε, γιατί χρειάζεται να μπορούμε να πετάξουμε προς όλες αυτές τις χώρες στον κόσμο. Να, να, να, να φαίνεται πως είμαστε ανοιχτοί και ότι ε, θα εξασφαλίσουμε όσο γίνεται καλύτερες υπηρεσίε. Εγώ είμαι πάντως σίγουρη ότι θα πετύχουμε, ότι θα πετύχουμε για τους κατανοητές και ότι ο κόσμος ε, σαν και εμένα, άνθρωποι σαν και δουλεύουμε μαζί με άλλους πολιτικούς, τις κυβερνήσεις και άλλους, ώστε να είναι όσο γίνεται πιο επιτυχής αυτή η διαδικασία. Και έπειτα, η Πρωθυπουργό ποτέ δεν μίλησε ούτε για απαλό ούτε για σκληρό Brexit. Είπε για Brexit. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε. Κύριε Βαντεκάμπο, δεν σας χρωστάω, δεν σας δίνω λογαριασμό, μου δείχνει το ρολόι. Και από τι δύο πλεόχθε λοιπόν του καναλιού τη μάχη θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη συμφωνία, δίκαιη διαπραγμάτευση και να εξασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να έχουν την επιλογή που είχαν εδώ και τόσο χρόνο. Σα ευχαριστώ. Παρακαλώ μην ξεπερνάτε με τι ερωτήσει σα ε, το χρόνο αγόρευσης. Θα πρέπει να μείνετε στα τρία λεπτά γιατί διαφορετικά θα χρειαστεί να κροτιάσουμε το τέλος της συζήτησης. Κυρία Μάισνερ. Κυρία Φώστερ, δεύτερη φορά παίρνετε το λόγο και μιλήσατε δύο φορές περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, και για τις παρουσιάσεις. Εγώ κυρίως ερωτήσεις θα κάνω. Βασικά τις εξή δύο. Ερώτηση πρώτη. Την επομένη του Brexit, αυτό που μάθαμε ε, ήταν ότι η αεροπλοεία θέλει να εξαιρεθεί από τον Brexit και τι διαπραγματεύσει. Ποιο από εσά συμμετείχε εκεί, ποιο το ζήτησε, ποιο το δήλωσε πού και τι σα απάντησαν. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Ε, γιατί αυτορά όλη την εναέρια κυκλοφορία που θα ε, θέλει να εξαιρείται. Ειδικέ ερωτήσει, κύριε Walsh, είπατε ότι θα θέλατε συμφωνία για την αεροπλοεία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου, που να είναι καλύτερο από Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και ε, όπως ε, είναι η συμφωνία με τον Καναδά. Και τι θέλετε να λέει αυτή η συμφωνία σε περίπτωση που διαπραγματευτούμε. Είπατε ότι ένα χρόνο πριν, κύριε ε, Κέννετη, πουλάτε τα εισιτήρια. Τι, τι πουλάτε ακριβώς ένα χρόνο πριν. Εγώ δεν αγοράζω το εισιτήριό μου για τις διακοπές ένα χρόνο πριν. Κύριε Ολύρη, είστε πολύ καλός ε, ε για συζήτηση και πολύ καλός διασκεδαστής και πάρα πολύ εφάνταστος και δημιουργικός και σας ερωτώ το εξής. Brexit ναι ή όχι. Εσείς τι θα κάνετε. Πόσο γρήγορα μπορείτε να καλύψετε το κενό εάν μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 δεν υπάρχει ασφαλές έδαφος και σίγουρη βάση. Σας φτάνει αυτό το διάστημα και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στο Open Sky. Λέτε πώς θα γίνει αυτό. Κύριε Κέννεντι, κυρίως ερώτηση για σας γιατί ε, πουλάτε ένα χρόνο πριν. Τι ποσοστό ακριβώς ένα χρόνο νωρίτερα για να καταλάβω τι θα σημάνει αυτό εάν κρατήσει αυτή η αβεβαιότητα ε, γιατί θα έχετε και πωλήσει μετά το χρόνο. Κύριε Κρόπ, σύντομα, γιατί είπατε ότι εμείς κάνουμε λάθος νόμους, εμείς νομοθετούμε μαζί με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνοι μας. Το λέω γιατί ε, αυτό είναι μια προσέγγιση που οδήγησε στο Brexit, γιατί πιστεύει ο κόσμος ότι όλα τα κακά έρχονται από τι Βρυξέλλες και όλα τα καλά από την πρωτεύουσά μου. Και σα ερωτώ, τι σημαίνει το Brexit για τη Lufthansa σε ε, αριθμούς. Και τέλος, κύριε Πασλάιτνερ, είπατε ότι 21 δισεκατομμύρια ε, θα χαθούν από τον τουρισμό. Αυτό φορά μόνο τη Μεγάλη Βρετανία, τι σημαίνει. Και το άλλο που είπατε, ότι γίνονται κρατήσει ένα με ένα μισή χρόνο πριν. Τι ποσοστό είναι αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μάισνερ. Ο κύριος Κράμερ από πλευρά των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Κύριε Κροπ, είπατε ότι χρειαζόμαστε δίκαιο εμπόριο. Έχετε απολύτω δίκαιο. αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δίκαιο εμπόριο. Έχουμε διαφορετικά τέλη, διαφορετικού αερολιμένε. Ακόμα για κάποιε εταιρείε έχουμε διαφορετικά τέλη στον ίδιο αερολιμένα. Αυτά μόνο δίκαια δεν είναι και σωστά. Και υπάρχει και ανταγωνισμό για τι μεγαλύτερε επιδοτήσει από τα αεροδρόμια. Με τον Brexit αυτό θα αλλάξει, θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα γίνει πιο δίκαιη η εμπορική αυτή συναλλαγή. Ryanair απαγορεύεται στη Δανία γιατί ε, αυτά που ισχύουν για τα κοινωνικά στη Δανία δεν θέλει να τα εφαρμόσει η Ryanair και σου λέει δεν πετάω καθόλου προκειμένου να τηρώ αυτές τις προδιαγραφές. Και για το Γιβραλτάρ παίζει σημαντικό ρόλο και κομβικό. Εδώ μας μπλοκάρει σε διάφορους ε, κανονισμούς και ρυθμίσεις για τα δικαιώματα ε, των επιβατών το Γιβραλτάρ. Μετά το Brexit τι θα γίνει θα έχουμε λιγότερα προβλήματα στην Ευρώπη όταν βγει το Γιβραλτάρ. Και ε, ένα τελευταίο που το έχω ξαναπεί. Ε, πολλά περιφερειακά αεροδρόμια είναι ελληματικά. Θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε από τον Καναδά που βάζουν τόσο υψηλά τέλη αεροδρομίου, ώστε να είναι κερδοφόρα όλα τα αεροδρόμια και να μην χρειάζεται να υποστηρίζονται από τον κρατικό προπολογισμό. Είναι αυτό ένα όραμα για το μέλλον. Γιατί το να πληρώνει ο μέσος φορολογούμενος άνδρας ή γυναίκα για όλους αυτούς του σούπερ μάνατζερ, μόνο κοινωνικό δεν είναι. ευχαριστώ κύριε Κράμερ, η κυρία Κλούν. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους σήμερα το απόγευμα. Ήταν μια πολύ θετική ακρόαση για τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη μετά από όλη αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα ερώτημα να θέσω, ένα γενικότερο ερώτημα. Κύριε Βόλς, μιλήσατε για τις ε, συμφωνίες για την αεροπορική μεταφορά. Χρειαζόμαστε παρεμφερείς συμφωνίες πιο ανοιχτές, με μεγαλύτερη ευελιξία, με την Ευρώπη των 27 και πράγματι. Έτσι έχουν τα πράγματα και αυτό θέλουμε. Προς όλους απευθύνω το ερώτημα ποια επικοινωνία είχατε με την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και με την ομάδα του κυρίου Μπαρνιέ εν ώψη της άφεξής σας εδώ σήμερα ε, με όλους αυτούς που παρακολουθούν και που βρίσκονται και εντός εθούσης και εκτός εθούσης. Έχετε να μας δώσετε κάποια νέα από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο επιδιώκει η πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, από ό,τι γνωρίζουμε δεν ε, το έχουν αυτό καθόλου συμπεριλάβει στο σκεπτικό τους ο Πρόεδρος. Από τους σοσιαλιστές θέλει κάποιο το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ο κύριος Μπαγιέ. Ευχαριστώ. Πράγματι θα βιαστώ, δεν θα μακρηγορήσω. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας. Για τις εξηγήσεις σας. Και εγώ εκφράζω τη λύπη μου για το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε άλλη επιλογή δυστυχώς. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύεται, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τελικά. Είπαμε ότι αν δεν υπάρχει πολιτική συνολική συμφωνία δεν υπάρχει καμία άλλη συμφωνία. Δεν συμφωνούμε με αυτό, δεν συμφωνούμε με την ε, καταληκτική προθεσμία του 2019. Θα λυθεί το θέμα αυξάνοντας απλά τα, την τιμή των εισιτηρίων ή υπάρχει άλλο τεχνικό ζήτημα. Η Ευρώπη έχει επενδύσει πολλά και στα περιφερειακά αεροδρόμια. Το σκληρό Brexit θα επηρεάσει αρνητικά τα περιφερειακά αεροδρόμια. Ίσως υπάρχει εξοικονόμηση του κόστου σε σχέση με τα τιμή του εισιτηρίου ξεκινώντας από περιφερειακά αεροδρόμια και όχι από κεντρικά. Και για τη Ryanair θα τροποποιήσετε την νομοθεσία για τις εταιρικές έδρες στην Ευρώπη ή για το πού θα γίνεται η κεφαλοποίηση της εταιρείας σας. Και με ένα ερώτημα για τον κύριο Ολύρη. Ολύρη, το Brexit θα επηρεάσει τη στρατηγική για τις διεπιρωτικές πτήσεις που θέλετε να ε, φτιάξετε και να δημιουργήσετε για τις εταιρείες low cost από την Ευρώπη προς τις άλλες επίρειες. Ευχαριστώ κυρία Γιούτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε σε σχέση με την, την απεσιοδοξία και την ε, τις, ε, τα φόβετρα που μας παρουσιάζει ο κύριος ε, Λύρη εγώ εμένα μου έρχεται να γελάσω, γιατί σε αυτά τα χαμηλά εισιτήρια ε, της Ryanair αφορούν ε, κακές πληρωμές, κακές αμοιβέ για τα πληρώματα και την επιλογή πολύ περιφερειακών αεροδρομίων. Και να, πρέπει να πω ότι είστε Ιρλανδοί και γι' αυτό και μετά το Brexit δεν θα έχετε προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ότι μετά το Brexit οι περισσότερες ε, ε, ε, ε, ιδιοκτησίες δεν θα είναι πια ευρωπαϊκές. Όλα αυτά οι εκφοβισμοί γιατί μας ε, τα παρουσιάζετε έτσι. Γιατί φοβάστε τι θα γίνει, ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα επιτραπεί στο Ηνωμένο Βασίλειο η πρόσβαση στους ανοιχτού ε, ουρανούς ή έχετε την ελπίδα ή τη βεβαιότητα ότι θα γίνει η αναθεώρηση του 868 του 2008 με αλλαγή της της οροφής του 48% ε, για τις εταιρείε τρίτων χωρών. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα ακολουθούν οι απαντήσει. Προτείνω με την αντίστροφη σειρά, μάλλον όχι, με την σειρά που μιλήσατε προηγουμένως, ο κύριος Γόλ πρώτος. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις σας. Θα ικανοποιείτε, έρχεται να ακούσετε ότι ο Μάικλ Ολύρη δεν έχει πάντα δίκιο και οι προβλέψεις του για τη κατάσταση μετά το Brexit δεν με βρίσκουν καθόλου σύμφωνο. Πιστεύω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει συνδεδεμένο με την υπόλοιπη Ευρώπη και η Ευρώπη των 27 θα παραμείνει συνδεδεμένη με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι προ όφελο και συμφέρον όλων των καταναλωτών και προ όφελο τη Ευρώπη πιστεύω. Ε, και είναι και προ το συμφέρον τη Ryanair δεν μπορεί να τα αναλάβει όλα η Ryanair να αντικαταστήσει όλα αυτά που θα εκλείψουν προς την Ευρώπη. Η EasyJet επίσης. Η αεροπορία ήταν μέγας ε, πρωταγωνιστής ε, στην ε, υλοποίηση και την επιτυχία της εσωτερικής αγοράς στους εθέρες. Αλλά χρειαζόμαστε ασφάλεια δικαίου, βεβαιότητα, το συντομότερο. Τα ίδια σχόλια κάναμε και προς τη Βρετανική κυβέρνηση. Αυτά που σας λέμε εδώ σήμερα. Η Βρετανική κυβέρνηση πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό το θέμα της αεροπορίας. Αυτό μπορεί να λυθεί με έναν τρόπο απλό και επικοδομητικό. Εγώ παραμένω αισιόδοξο ότι θα λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και η Ryanair θα συνεχίζει να πετάει από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Πόσο και αν θαυμάζω το Μάικλ Λύρη, διαφωνώ ε, εντόνως μαζί του. Επίσης, οι υποδομές που έχουν στηθεί πριν από πολλά χρόνια για να αντιμετωπιστούν τα θέματα της ιδιοκτησίας και του ελέγχου και που ε, αφισβητούνται, θα παραμείνουν ισχύ. Είναι απαραίτητε οι δομέ και οι υποδομέ και ελπίζω να μην χρειαστεί να ε, τις αντικαταστήσουμε κάπου αλλού. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, εμείς ως IAG θα συνεχίσουμε να τηρούμε όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς και ελπίζω να βρεθεί ένας τρόπος να παραμείνει ο σημαντικός συνεισφορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ευεργέτης ε, των, ε, του έργου της ΕΑΣΑ. Είναι σημαντικό αυτό. Ο, ο Οργανισμός Ασφάλειας ε, στις αερομεταφορές ε, είχε σημαντική συνεισφορά και ρόλο και στην Ευρώπη των 27 και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Επειδή έχω περάσει μια ζωή ολόκληρη στην αεροπορία, ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ κύριε Βόλς που τήρησατε και το τρίλεπτο. Ο κύριος Ολύρη. Εγώ θέλω να απαντήσω με ένα, σε δύο ε, ότι οι διμερείς δεν θα είναι ε, λέει, ε, επιλογή γιατί κανένας από τους 27 δεν θα θελήσει να διαπραγματευτεί διμερή συμφωνία. Οι 27 θα ενωθούν. Οι Βρετανοί θα χρειαστούν θεωρήσεις για να έρθουν στην Ευρώπη. Ναι, θα χρειαστούν, αλλά μην ανησυχείτε γιατί θα υπάρχουν πτήσεις μετά το Brexit ανάμεσα στον Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βρετανία, την Ευρώπη, ούτε με το Ιρλανδία. Και ούτε μπορείτε να μας πείσετε κυρία Φώστερ ότι όλα ωραία και καλά θα πάνε γιατί θα υπάρξει συμφωνία. Δεν υπάρχει μηχανισμός στην Ηνωμένο Βασίλειο για να υπάρξει συμφωνία. Δεν ξέρουν τι θα πει συμφωνία, δεν ξέρουν ούτε καν τι θέλουν εκτός από το να φύγουν από τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτά είναι δικό σας υπόθεση, δικό σας κόμμα. Σας προτείνω να μιλήσετε μαζί του. Γιατί η Γερμανίδα, κυρία, δεν θα υπάρξει δική μεταχείριση για την αεροπλοή. Μην νομίζετε ότι εγώ το παίρνω ελαφρά το Brexit. Πιστεύω ότι το Brexit είναι ε, μεγάλο μπάχαλο. Η Βρετανία θα υποφέρει, η Ευρώπη θα υποφέρει, θα έχουμε αντική μεγέθυνση, θα είναι χάλια για τον κλάδο μας, αλλά Εμεί, επειδή μπορούμε να πάρουμε τα αεροπλανάκια μας από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούμε να γλιτώσουμε λίγο. Αλλά κατά τα άλλα μην νομίζετε ότι το παίρνουν ελαφριά. Οι Βρετανοί θα καταλάβουν πάρα πολύ καλά ότι δεν θέλουν να πάνε ούτε στην Ιρλανδία ούτε στη Σκωτία για διακοπές και τότε θα συνέλθουν ξαφνικά. Κύριε Κρέμερα, σα αγαπώ, αλλά πραγματικά ε, τρέφεται πάντα. Όχι μόνο πάμε στη Δανία, είμαστε η μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη εταιρεία στη Δανία. Είμαστε νούμερο 3 στην Κοπενχάγη μέσα σε 18 μήνε. Επίση έχουμε 100% την ανάπτυξη τη Κοπενχάγης τα τελευταία δύο χρόνια. Τώρα, γιατί εμείς δεν ε, αφήνουμε τα σκάφη μας εκεί στη Δανία, υπάρχει ένα παράξενο μοντέλο που επιτρέπει στη, στην, ε, στα συνδικάτα της ΣΑΣ να μπλοκάρουν τα δικά μας αεροπλάνα παρότι τα δικά τα πληρώματα και οι δικοί μας επιβάτες δεν το θέλουν, όμως από τη στιγμή που η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα σε σχέση με αυτόν τον συνδικαλιστικό, τη συνδικαλιστική τρομοκρατία, τότε δική σας ντροπή είναι αυτό και όχι δική μας τώρα για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Βρετανική κυβέρνηση. Ε, δεν λυπούμε, αλλά ξαναλέω ότι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι κάνουν όταν τους ρωτήσεις πώς θα τα καταφέρουν αυτά εκεί δεν έχουν ιδέα. Ανοιχτή ουρανή ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη νομίζω ότι είναι συμφωνία με το Πακιστάν. Σίγουρα πολλοί Πακιστανοί θα θέλουν να έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι πολλοί Βρετανοί θέλουν να πάνε στο Καράτσι για διακοπέ. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν θα υπάρχει συμφωνία, δεν θα υπάρχουν πτήσει. Δεν υπάρχει νομικό μηχανισμό σύμφωνα με τον οποίο να μπορεί να λειτουργήσουν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε σε περίπτωση hard Brexit. Δηλαδή δεν έχει νόημα να έχουμε ψηλότερε τιμέ σε κάποια αεροδρόμια σε κάποιες αεροπορικέ εταιρείες προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Είτε θα υπάρξουν ανοιχτοί ουρανοί, είτε διμερείς συμφωνίες. Αν δεν υπάρξει το ένα ούτε το άλλο, δεν θα υπάρξουν πτήσεις για μέρες και εβδομάδες. Επίσης, Έχουμε πολύ καλές αμοιβέ ε, στη Ryanair. Γύρω στους 5.000 πιλότες έχουμε σε λίστα αναμονής που θέλουν να πιάσουν δουλειά σε εμά και από την Αλτάλια και από την British Airways όπου υπάρχουν χαμηλότερα στάνταρ ε, στις υποτιθέμενες ε, παλιές εταιρείε και στις εθνικρατικές εταιρείε, Το 20% των μετόχων μας είναι Βρετανοί. Εμείς έχουμε διαρκώς μερίσματα και αν οι Βρετανοί μέτοχοι χρειαστεί να πουλήσουν, αναγκαστούν να πουλήσουν, θα του τα αγοράσω εγώ ξανά. Ανοιχτή πρόσβαση. Ελπίζω πω το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιστρέψει την απόφαση για τον Brexit και όταν το Σεπτέμβριο του 2018 θα διαπιστώσουν ότι δεν θα υπάρξουν πτήσει προ την Ισπανία, την Πορτογαλία και ούτε και την Ιταλία, το για το καλοκαίρι του 2019, ο μέσο Βρετανό ψηφοφόρο που δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, ε, ε, θα δεν καταλαβαίνει ούτε τη τόμα, αλλά καταλαβαίνει ότι θέλει να πάει φτηνές διακοπές στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα και στην Ισπανία, θα καταλάβει πως παραπλανήθηκε ε, με το δημοψήφισμα του Brexit πέρυσι και θα αλλάξει τη γνώμη του. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύω πως οι Βρετανοί θα αλλάξουν την γνώμη τους, γιατί διαφορετικά ε, θα περάσουν πολύ πολύ δύσκολα τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ολύρη. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κρόπ. Α, συγγνώμη, ο κύριος Κένετη πρώτα. Θα, αναφερθώ, θα αναφερόμουν σε αυτό που είπε ο κύριος Κάμπ. Τι συμβαίνει με τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες. Εάν υπάρξει ε, σκληρό Brexit και την πρώτη ημέρα ε, μετά δεν υπάρχει συμφωνία, θα πάμε στις διμερείς πριν από το 73 είχαν συγγραφεί στη δεκαετία του 40, του 50 και του 60 και προσδιορίζουν ποιες είναι οι αεροπορικές εταιρείες που μπορούν να εξυπηρετούν την αγορά. Άρα ε, πολλές από τις εταιρείες που βλέπετε εδώ δεν υπήρχαν τότε και δεν θα έχουν δικαίωμα να πετούν. Θα είναι λιγότερες οι επιλογές για τους πολίτες και τότε οι πτήσει ήταν πολύ λιγότερες και άρα οι επιλογές των καταναλωτών θα είναι πολύ λιγότερες. Από εκεί και πέρα από αμερικανικής πλευράς τα joint ventures που έχουμε με την KLM, με την British Airways, με τη Lufthansa κτλ. Λίγουν, ολοκληρώνονται και το νομικό θεμέλιο, τα νομικά στοιχεία φαντα... υποθέτουν ότι υπάρχει κοινός ενεάριος χώρος. Δηλαδή εγώ πέταξα από τη ΣΥΠΑ στη Φραγκφούρτη και ήρθα μετά στις Βρυξέλλες. Αν πετάξω στο ε, ε, Χήθρο και πάω μετά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αυτό είναι συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ε, υπόλοιπη Ευρώπης για να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία μετάβαση των επιβατών. Όταν σας είπα ότι το 50% της κυκλοφορίας του Χήθρου πηγαίνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό γίνεται λόγω των joint ventures, των κοινών συμπράξεων, οι οποίες θα λήξουν από την πρώτη μέρα του σκληρού Brexit. Και έχουμε τα μικρά και μεσαία αεροδρόμια. Από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση από αμερικανικές πόλεις σε μικρά περιφερειακά αεροδρόμια. Έχουμε ένα σύστημα με hub, ε, στέλνουμε την κίνηση στο Heathrow και εκεί αλλάζουν μέσω joint venture ε, ετεροπορική εταιρεία και ο Αμερικανός τουρίστα τουρίστας, ή επιχειρηματίες έτσι φτάνει σε περιφερειακό αεροδρόμιο σε μικρότερη κοινότητα. Εμείς θεωρούμε ότι ο αντίκτυπος θα είναι πολύ μεγάλος, ιδίως από την αμερικανική πλευρά γιατί θα είναι εξαιρετικά πιο δύσκολο να μεταφερθούν οι Αμερικανοί σε αυτά τα μέρη, τα μικρά και τα περιφερειακά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας Κρόπ έχει το λόγο. είναι ένα σχόλιο. Στον Αμερικανό προλαλήσαντα. Αν κάνουμε νέα διαπραγμάτευση, θα επιθυμούσαμε και εμείς το αυτό όπως θέλετε εσείς από το Χήθρο να πετάτε στην υπηρετική Ευρώπη, θα θέλαμε και εμείς από τη Νέα Υόρκη στο Σικάγο. Το ίδιο ισχύει για τον έλεγχο και την ιδιοκτησία. 75% δεν είναι America First, ε, λένε ε, προτιμησιακό καθεστώς για αμερικανικές εταιρείες. Εμάς είναι 50%. Άμα λέτε 75% είναι πρόβλημα. Πάω στις ερωτήσεις για τον κύριο Φάντεμ Κάμπ. Αν έχει αυτό επιπτώσει στους ναύλους. Καταρχάς, ελπίζω να το είχα πει, ότι ε, θέλουμε να έχουμε μια αρρύθμιση τελικά και πολλά να μην αλλάξουν. Η Ευρώπη είναι γεμάτη ε, από ε, point to point carriers. Έχουμε την Norwegian που πετάνε στην Ευρώπη γιατί είναι στον νεόχη Νορβηγία. Έχουμε και άλλους αερομεταφορείς. Wizz Air στην Ανατολική Ευρώπη, Eurowings που είναι της δικής μας, ε, της ε, Lufthansa, Transavia από τον Όμιλο Air France KLM. Και η Ryanair από ό,τι άκουσα μπορεί να κινείται όπως θέλει ελεύθερα στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Η Jacqueline Foster είπε για την παράλληλη συζήτηση που γίνεται για νέες ρυθμίσεις για δίκαιο ανταγωνισμό. Αυτό δεν είναι προστατευτισμός, το υπενήχθη εγώ, αλλά πρόκειται για εταιρείε που δεν έχουν σχέση με το Brexit, αλλά στον περσικό κόλπο έχουμε μικρές χώρες με τεράστιο στόλο. Αεροσκάφη ούτε δικαίωμα στην απεργία έχουν ούτε τίποτα από τις δικές μας ρυθμίσεις και με αυτούς εμείς πρέπει να ανταγωνιζόμαστε. Και θέλουμε και ίσους κανόνους παιχνιδιού. Ε, δεν είμαστε στον ΠΟΕ η αεροπορία. Οι περισσότεροι δεν το ξέρουν αυτό. Και εμείς εξαρτώμαστε από κάθε εκατοστό της συμφωνίας ε, ή των συμφωνιών η αυτοκινητοβιομηχανία και κάποιοι άλλοι που συμπεριλαμβάνονται στον ΠΟΕ έχουν περιθώριο χειρισμών. Εμείς όχι. Η κυρία Μάισνερ είπε ότι είπα εγώ ότι βγάζετε λάθος νόμους. Μπορεί να το είπα κατά λάθο. Εννοούσα ότι έχουμε νόμους που μπορεί να μην τους αγαπάμε όλοι, αλλά θα πρέπει να τους εφαρμόζουμε. Και στην εσωτερική αγορά Υπάρχουν ε, νόμοι που σωστά ψηφίζονται με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να τους εφαρμόζουμε. Δεν λέω ότι είναι σωστή η νόμη ή λάθο. απλώς θα πρέπει να του εφαρμόζουμε και έχουν κάποιες επιπτώσεις και οικονομικές. Ο κύριος Κράμερ τόνισε το θέμα του δίκαιου εμπορίου και ανταγωνισμού. Εμείς Έχουμε πρόβλημα. Αν θέλουμε να πουλήσουμε ε, φθηνότερα εισιτήρια, δεν μειώνεται ούτε η κυροζήνη, η τιμή της, ούτε τα τέλη αερολιμένων. Υπάρχουν αεροδρόμια που κάνουν εκπτώσεις 50% για όλους εκτός από τους βασικούς πελάτες. Ε, και αυτό μας πλήττει εμάς. Εμείς έχουμε 100.000 εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν όλα να είναι στην πλάτη των εργαζομένων. Ε, τα εισιτήρια για να πέσουν θα πρέπει να μπορεί να ζει ένας εργαζόμενος ε, στη Λούφθανζα από το μισθό που παίρνει. Και προς το παρόν αυτό ισχύει. Και θα ε, θέλουμε να ε, αγωνιστούμε, να ανταγωνιστούμε ελεύθερα και δίκαια για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάστλαϊτνερ, τελευταίος. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Για, το, για τα θέματα των θεωρήσεων, το εξετάζουμε από την πλευρά της κινητικότητας του προσωπικού του Ηνωμένου Βασίλειου. Θα χρειαστούν θεωρήσεις όταν θα τους αποσπάσουμε σε διάφορα άλλα μέλη στην Ευρώπη για να εξυπηρετήσουν τους προορισμούς που εμείς παρέχουμε στους πελάτες μας. Αυτό ε, κοιτάμε τώρα. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο, η ερώτηση. Συμφωνώ μαζί σας, απαντά ο κύριος Πασλάιτνερ. Εμείς το εξετάζουμε από την οικονομική σκοπιά και τα θέματα του προσωπικού μας, αλλά και από πλευράς τουρισμού είναι πολιτική διαδικασία. Αν θέλετε διαδικασία ε, fast track για ορισμένες χώρες, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Δεν, δεν μπορώ να το σχολιάσω εγώ. Ε, εμείς θα κάνουμε αξιολόγηση κυρίως για το οικονομικό σκέλος, για την οικονομική πτυχή του θέματος. κυρία Μάισνερ. Το ερώτημα για τις ενδεχόμενες απώλειες. Αναθέσαμε μια μελέτη και προέκυψε μια απώλεια 21 δις ε, στον τουρισμό στα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης. Από το γεγονός ότι δεν θα στέλνει τουρίστες στο Ηνωμένο Βασίλειο στους υπόλοιπους 27, 21 δις. Σε αυτό αναφερόμαστε. Uh, και το θέμα των κρατήσεων δεν είναι ότι οι τουρίστες, οι δικοί μας πελάτες κλείνουν 1,5 χρόνο πριν τις διακοπές τους, παρόλο που όλο και νωρίτερα. Αλλά εμείς κοιτάμε τις δυνατότητες, τα δρομολόγια, ε, τους προορισμούς, τις κλίνες, τα ξενοδοχεία, οι tour operators. 12 ε, με 18 μήνες πριν κάνουν τον προγραμματισμό τους. Ευχαριστώ πολύ. Πριν φύγετε, θα ακούσουμε και την εκπρόσωπο της ΕΡΒΑΣ και θα ξαναδώσω το λόγο για ένα λεπτό σε όλους σας. Έχω την ιδιαίτερη τιμή να καλωσορίζω την Αταλία Γάχ που εκπροσωπεί την Airbus και όπως όλος ο κόσμος έχετε τον ίδιο χρόνο. 5 με 7 λεπτά, παρακαλώ. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμπληρώσω την εικόνα που σας ήδη παρουσίασαν οι πελάτες μας που είναι τα αεροπορικές εταιρείες. Η Airbus λοιπόν χρησιμοποιείται συχνά ως σύμβολο επιτυχίας ε, επιχειρηματικής ολοκλήρωσης και ενοποίησης γιατί εμείς καταλαμβάνουμε το 5% της παγκόσμιας αγοράς κατασκευής αεροσκαφών μπορέσαμε να αναπτυχθούμε, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να δημιουργήσουμε καινοτομία και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Όμως πρέπει κανείς να κατανοήσει το επιχειρηματικό μοντέλο. Τα ε, πτερίγια φτιάχνονται στον Ηνωμένο Βασίλειο, η άτρακτο στη Γερμανία, το ρίγχος και βασικά ε, τεχνολογικά εξαρτήματα στη Γαλλία ε, και σε άλλες χώρες βεβαίως άλλα πράγματα. Ο, έχουμε παγκόσμια επιτυχία και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στην ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και ε, αγαθών, εμπορευμάτων που κυκλοφορούν και ταξιδεύουν και διαμετακομίζονται αντιστοίχως απρόσκοπτα. Από τη μία χώρα στην άλλη. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να έχουμε κατοχήρωση των θέσεων, κατοχήρωση απασχόλησης. Εάν τώρα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σίγουρα είναι μια χώρα που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κατασκευαστικό μας αποτύπωμα. Όλα τα φτερά ε, των αεροσκαφών κατασκευάζονται στην Νότιο Ουαλία και χωρίς, την, χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή το Airbus θα είναι μόνο bus, θα είναι μόνο λεωφορείο και όχι ε, ένα αέριο αεροσκάφος, εν πάση Airbus. Έχουμε πάρα πολλούς προμηθευτές και ε, λοιπές εταιρείε με τις οποίες συνεργαζόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, άρα πολύ μεγάλη συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, με πανεπιστήμια. Ε, όλα αυτά διασχίζουν τη μάχη επανειλημμένος. Δηλαδή 80.000 φορές διασχίζουμε τη μάχη ετησίως και τίθεται το ερώτημα τι θα συμβεί με το Brexit. Ξέρετε ότι η Airbus δημόσια άσκησε λόμπι και άσκησε πίεση κατά του Brexit κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος, όχι για λόγους ιδεολογίας, αλλά γιατί ήταν βασική επιχειρηματική κοινή λογική. Εμείς είμαστε ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο στερέωμα. Η ανταγωνιστικότητα των διαφόρων εργοστασίων μας και κέντρων μας σε όλη την Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική. Σκοπός μας είναι, είναι να ανταγωνιστούμε την Κίνα και πρέπει να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε ε, όλα τα κεκτημένα μας. Έχω πέντε λεπτά στη διάθεσή μου και θα ήθελα να αναφέρω τα βασικά μηνύματα. Ε, έχουμε περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις, γιατί ξέρουμε τελικά ποια μορφή θα λάβει το Brexit. Το βασικό είναι η κινητικότητα των εργαζομένων πρέπει γρήγορα να φέρουμε ανθρώπους, να τους αποσπάσουμε στα διάφορα εργοστάσια. Πώς μπορεί ένας εμπειρογνώμονας, ένας ειδικό που είναι απασχολούμενος στο Ηνωμένο Βασίλειο να μεταφερθεί γρήγορα. Έχουμε προμηθευτές της Rolls Royce για τους κινητήρες. Πώς θα μεταφερθούν αν υπάρχει πρόβλημα και πώς θα διασχίσουν τη μάχη. Πρέπει να το κάνουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Άρα αυτό είναι το βασικό. Ένα πρώτο στοιχείο πέρα από τους 1.900 ανθρώπους που είτε είναι Βρετανοί που έχουν αποσπαστεί και μόνιμα είναι κάτοικοι ε, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εργάζονται για μας εκεί ή 1.900 επίσης Ευρωπαίους που έχουν αποσπαστεί και εργάζονται και μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές είναι οι βασικές μας ανησυχίες. Μετά έχουμε τους ελέγχους στα σύνορα και τις κανονιστικές αποκλήσεις στην νομοθεσία των διαφόρων χωρών. Διάφορα εξαρτήματα, διάφορα ανταλλακτικά τα στέλνουμε και τα λαμβάνουμε από διάφορες χώρες. Επομένως μας ενδιαφέρει να μην υπάρχουν δασμοί και να μην περνάμε από το ελωνίο από αυτή την έννοια, με καταβάλλοντας δασμούς. Και Υπάρχουν κάποιες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα υπάρχει λύση σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου. Θα υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο ΠΟΕ στην οποία θα μπορούσαμε να βασιστούμε για να ελαφρυθούμε από την καταβολή των δασμών. Εμάς μας ενδιαφέρει επίσης και ο αντίκτυπος που, αντίκτυπος που δεν έχει να κάνει με το δασμολογικό κόστος γιατί η έλεγχη στα σύνορα είναι προβληματική ακόμα και αν είναι αδεσμολόγητα τα προϊόντα. Γιατί σημαίνει ότι ε, χάνεται χρόνος. Φαντάζεστε φτερά αεροσκαφό να παραμένουν στα σύνορα και να μην μπορούν να τα παραλάβουμε, να μην μπορούμε να, ε, ε, να εκπληρώσουμε τις προθεσμίες που έχουμε ε, υποσχεθεί στους πελάτες μας. Και αν υπάρξει και συμφωνία τελωνιακή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν κάτι τέτοιο συμβεί, παραμένουν ζητήματα με τους ελέγχους στα σύνορα, με τους κανονισμούς. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι έλεγχοι θα διενεργούνται αποτελεσματικά. Είναι ένα θέμα στο πάνω στο οποίο χρειάζεται δουλειά. Ήδη Μιλήσαμε για την ΕΑΣΑ και τη σημασία που έχει για το δικό μας κλάδο. Δεν θέλουμε αποκλήσεις προφανώς σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς για την ασφάλεια, για την πιστοποίηση. Άρα θα πρέπει να έχει ευελιξία και η άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι το θέμα μόνο η σύγκληση της κανονιστικής νομοθεσίας, αλλά να υπάρχει και ένας μηχανισμός θέσης σε ισχύ, υποχρέωσης, επιβολής των κανόνων, που να πηγαίνουν ε, χέρι-χέρι αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να έχει κανείς το ένα και να μην έχει το άλλο. Συμμόρφωση, δηλαδή, χωρίς μηχανισμό επιβολής των κανόνων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ανταγωνιστικότητας και υπάρχει και το θέμα, ένα τρίτο θέμα ε, που είναι οι πτυχές της εταιρικής σχέσης. Έχουμε θυγατρική για τα θέματα τα διαστημικά με το Γαλιλαίο που δίνει εξαρτήματα στη Γερμανία και έχουμε θυγατρική που εδράζεται στο Αμένο Βασίλειο. Ε, θα τελειώσει αυτή η συνεργασία, τι θα γίνει. Έχουμε το ΣΕΖΑΡ, τους καθαρούς ουρανούς. Πώς θα συνεχιστούν αυτές οι εταιρικέ σχέσεις. Εμείς θέλουμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να τις διασφαλίσουμε, να τις εξασφαλίσουμε, να μπορέσουν να συνεχιστούν. Με δύο λόγια λοιπόν, χρειαζόμαστε συμφωνία, θα είναι δεινή η θέση μας χωρίς συμφωνία, παραμένει αβεβαιότητα για τις συγκεκριμένες πτυχές της συμφωνίας και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια σκακέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άρα. Συζήτηση. Ένα λεπτό έκαστος για να κάνετε την ερώτησή σας. Και θα είμαι αμήλικτη. Κύριε Μπαχ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω την ερώτησή μου στα γερμανικά η αεροπορία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την εμπιστοσύνη, κυρίως των πελατών. Και έχω την εξή ερώτηση. Εσείς προσπαθήσατε να εκπέμψετε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ακόμα και ο μεγαλύτερος ε, αισιόδοξο κλονίζεται και ε, το Μάρτιο του 2019 δεν μπορεί να τηρηθεί ως προθεσμία. Δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία μέχρι τότε. Ρωτώ λοιπόν, σίγουρα για να ε, εγγυηθείτε αυτή την εμπιστοσύνη πρέπει να εξασφαλιστείτε κάπως. Πώς θα εξασφαλιστείτε. Σας ασφαλίζουν ασφαλιστικές εταιρείες. Μήπως αυτές ε, θα είναι οι κερδισμένοι από το Brexit. Κύριε Ρικέ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις σκέψεις έχω να κάνω, τρία σχόλια έχοντας ακούσει όλους τους ομιλητές. Πρώτον, είπαν οι ομιλητές από τα αεροδρόμια ότι το Brexit μπορεί να θεωρείται ως πολιτική υπόθεση. Ε, ατυχήσαμε όμως. Είναι πολιτική απόφαση και η οικονομία είναι θύμα της πολιτικής. Ακούγοντας όλο το πάνελ, εγώ διακρίνω κάποιο πανικό. Κανένας δεν έχει σαφή εικόνα ούτε τι μελιγενέστε, ούτε τι λύσεις μπορούμε να προτείνουμε. Δεύτερο σχόλιο. Θα παραθέσω την Πρωθυπουργό Τερέζα Μέη. Το Brexit είναι Brexit. Τι άλλο μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να είναι ο λίγον Brexit, ε, μια άλλη διαφορετική πολιτική πρόταση. Και στην Ευρώπη έχουμε την καλή συνήθεια να λέμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία γιατί τίποτα δεν συμφωνηθούν τα πάντα. Συμπέρασμα λοιπόν. Αναγκαστικά. Πού είναι αυτοί που είναι υπέρ του Brexit. Εγώ δεν έχω συναντήσει κανέναν πάντως. Ε, αναγκαστικά λοιπόν πάμε κατευθείαν στον κρεμό. Από ό,τι άκουσα και είμαστε και πολύ κοντά. Ευχαριστώ η κυρία Άντερσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Να σας πω ότι εμείς είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλω να σας ρωτήσω ειδικά ποιος ήταν ο αντίκτυπος στην έρευνα και στην ανάπτυξη όσον αφορά τα προγράμματα χρηματοδότησης. Και επίσης όσον αφορά το αρμονικό πλαίσιο σχέσεων, ε, επιτροπές κοινωνικού διαλόγου και τον τρόπο με τον οποίο τώρα λειτουργούν όλα αυτά υπέρ όλων, δηλαδή τόσο υπέρ των εργαζομένων και συνδικάτων τους όσο και εργοδοτών. Και έπειτα ευρύτερα, τι κάνετε με τους ε, εκπατρισμένους σας και την ελευθερία ε, κυκλοφορίας των ατόμων. Είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά το χειρισμό από πλευρά τη Ιταλική κυβέρνηση τη κατάσταση και το γεγονό ότι δεν θα προστατευτούν ισότιμα οι πολίτε. Υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά την επανένωση οικογενειών και βέβαια ε, το πρόσχημα αυτό που χρησιμοποιείται ότι η μετανάστευση κάθε είδου ε, ε, υποφέρουν από αυτά τα προσχήματα. Υπάρχει τεράστια αύξηση ρατσισμού και Ε, Πώ επηρεάζει αυτό το δικό σα εργατικό δυναμικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άντερσον και κλείνουμε με τον κύριο Γκίλερ. Γκίλερ. Γκάλερ. Γκάλερ στα γερμανικά, όχι και πολύ. Α, γκαλέρ, ναι, γαλέρα. Ε, λοιπόν, έχω μια ερώτηση προς την κυρία Ερά, ε, την οποία άκουσα προσεκτικά. Και αναγκαστικά βγάζω το συμπέρασμα ότι αν είναι τόσο δύσκολο ή τόσο αβέβαιο όλο αυτό που θα συμβεί, αν μπορεί να διατηρηθεί η αλυσίδα παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν είναι τόσο αβέβαια η κατάσταση, αν πραγματικά μπορούν να κυκλοφορούν οι εργαζόμενοι, τότε λογικό συμπέρασμα θα πρέπει να είναι να παράγεται ε, το προϊόν στην υπηρετική Ευρώπη. Το έχει σκεφτεί αυτό η Airbus. Ευχαριστώ. Στρέφομαι και πάλι προς την κυρία Ερά για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Έρευνα και ανάπτυξη. Και... Πολύ σημαντικά αυτά που ρωτήσατε και θα σας ζητήσω σε όλους είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά θέλουμε να κλείσουμε με ένα λεπτό. Τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε, αν έπρεπε να κλείσετε. Αγαπητοί οικονομικοί φορείς, το ξέρω πως είναι δύσκολο, ταυτόχρονα μας επιτρέπει εμάς να ακούσουμε ακριβώς το ζουμί. Έχετε το λόγο. Είναι δύσκολο να σχολιάσουμε τι θα συμβεί όσον αφορά την έρευνα καθώς και, τους, ε, και με τους εκπατρισμένους μας ε, ε, πολίτες. Χρειάζεται συμφωνία πρώτα. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πού θα βασιστεί η διαπραγμάτευση, είναι δύσκολο να σχολιάσουμε. Κανονικά θα μπορούσε κανείς να καταλάβει πού θα έπρεπε να εστιάσει, αν ήταν κομμάτι του ορίζον 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά όπως θυμήσαμε υπάρχει αυτή η κειμενόμενη διάσταση όπου τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι ότου όλα συμφωνηθούν. Δεν ξέρουμε καθόλου μα καθόλου ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Είναι όλα πολύ ρευστά. Δεν μπορώ να σχολιάσω ε, ποια θα είναι η τελική πρόταση του Ηνωμένου Βασίλειου για τους, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα μόλις ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις βεβαίως κοιτάμε και άλλους και κοινά project και νομίζω πως το πολιτικό ζήτημα ε, είναι βασικό οι πολιτικοί πρέπει να βρουν κάποια συμφωνία για το πώς θα λύσουμε το θέμα αυτό, γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε όλοι ε, ενώπιον προβλημάτων. Το άλλο θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα και πώς θα μπορέσουμε γρήγορα να αλλάξουμε τις δραστηριότητέ μας, πώς θα μετακινήσουμε τις δραστηριότητε μας στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, στην ε, Πυρωτική Ευρώπη. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το πολιτικό αποτέλεσμα. Βεβαίω θα κοιτάξουμε, θα εξετάσουμε τη μακροπρόθεσμή μας ανταγωνιστικότητα στα διάφορα μας εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά θέλω να τονίσω την τεχνογνωσία αλλά και τα, τις εγκαταστάσεις και όλα τα, τα ατού. Εμείς δεν αγωνιζόμαστε κατά το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι. Εμείς ε, θεωρούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη βιομηχανία είναι ένα από τα καλύτερα κράτη στον κόσμο. Αλλά τα θέματα που προκύπτουν από τον Brexit είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας αλλά πιθανότατα είναι πολύ πιο σημαντικά για την ολόκληρη την ασυλισίδα ε, προμήθειών που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί ξέρετε υπάρχουν επενδύσεις στα συστήματα IT όπου πρέπει κανείς να μπορεί να προσαρμόσει τις διαδικασίες, αλλά πραγματικά η... τα τελωνία, οι ρυθμίσεις αλλάξουν ώστε να υπάρξει διαταραχή στην ροή παραγωγής, Βεβαίω οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις θα είναι αυτές που θα υποφέρουν περισσότερο. Και αυτό είναι προβληματισμός μας και ανησυχία μας, ειδικά αν είναι χαμηλά η λίρα. Χαμηλά, όπως είπαμε, και οι δοκιμάσει στις τιμές αυτές μπορεί να είναι πολύ σημαντικές για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ευχαριστώ. Κυρία Έρχαρτε, αν είχατε να μου πείτε ένα μικρό μήνυμα, ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε. Το μήνυμα είναι ε, είναι ότι το να μέναμε ήταν καλύτερα, το να φύγει κανείς σημαίνει ότι ε, έχετε μόνος του στον κόσμο, αλλά από την άποψη την επιχειρηματική είναι αυτή η, η άποψη. Τώρα όμως η πολιτική είναι υπεύθυνη. Α ελπίσουμε ότι θα βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για την ευρωπαϊκή μεταπητική βιομηχανία και για τους πελάτες μας, τις αεροπορικέ εταιρείε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Έρχερ. και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκόλτενερ. Κύριε Πρόεδρε, για τα που είναι στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ενιαία αγορά, το βασικό θέμα είναι θα είναι ποιε θα είναι οι αρχέ εξόδου ε, για αυτέ τι εταιρείε που θα βγουν από τον ευρωπαϊκό ενιαίο χώρο και ποιοι θα είναι οι όροι πρόσβαση στην ενιαία αγορά για αυτού του ε, φορεί. Ε, γιατί υπάρχουν τώρα μοντέλα και μπορούν να αντικατασταθούν. Ευχαριστώ κύριε Γκόλντενέλ. Ο κύριος Τόλαντ. Η Ιρλανδία είναι η πιο εκτεθειμένη χώρα λόγω συνδυσιμότητας μετά το Brexit. Θα πρέπει να θυμηθούμε αυτό που είναι κλειδί, ότι τους λείπει η ε, συνδυσιμότητα μέσα στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Για την ΕΚΑΚ πιστεύω πως είναι ένας κρίσιμος ακρογωνίος λίθος και θα πρέπει να επικρατήσει κοινή λογική. Ε, δεν είναι θέμα απόλυτη συμφωνία με τις κυρίες Φώστερ και τις παρατηρήσεις της και έπειτα ότι χρειάζεται σαφήνεια όσο γίνεται πιο σύντομα. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν υπάρχει σαφήνεια αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Walsh, ένα λεπτό. Τι μήνυμα έχετε να μας δώσετε. Ευχαριστώ. Η αεροπλοή είναι μια από τις επιτυχημένες ιστορίες τη Ευρωπαϊκής Ένωση και με χαρά λέω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ανέκαθεν στήριζε ανοιχτό, ελεύθερο, ελεύθερη και απορριθμισμένη αγορά αερομεταφορών. Η Ευρώπη σπρώχνει μια ανοιχτή πόρτα. Χρειάζεται να δουλέψουμε ώστε να συμφωνήσουμε σε μια καθολική συμφωνία αερομεταφορών ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση που θα διατηρεί όλα τα ωφέλη για τους καταναλωτές που έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα και παραμένω αισιόδοξο ότι θα το καταφέρουμε αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Ολύρη. Εγώ με την, έχω την αντίθετη απόψη. Πιστεύω πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αλλάξει την πολιτική της, οδεύει προς ένα σκληρό Brexit, που δηλαδή πάυση πτήσεων όλων των πτήσεων ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη από τον Απρίλιο του 2019 και μετά. Ε, η προθεσμία δεν είναι ο Μάρτιος του 19, η προθεσμία είναι ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018. Τότε θα αρχίσουμε να ακυρώνουμε τις πτήσεις έξι μήνες πριν από το Μάρτιο του 19. Δεν θα περιμένουμε. Ε, το Μάρτιο του 19. Και τελευταία μου παρατήρηση κάποια σχόλια από τον κύριο Κρέμερ για το ότι θα χάσουν τα περιφερειακά αεροδρόμια λεφτά. Να σας πω πώς θα πάψουν να, χάσουν, να χάνουν λεφτά. Το Σαρλερουά έχει 20.000 ε, επιβάτες ε, το χρόνο και έχανε λεφτά. Τώρα έχει πάει στα 29 εκατομμύρια επιβάτες και κερδίζει λεφτά. Ο κύριος Κέννεντι εγώ έχω πάει σε πολλά μέρη, σε πολλές χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Πολλοί βλέπουν την αεροπλοεία ως τις άλλους κλάδους και, βλέπουν, και λένε δεν θέλουμε να συζητήσουμε τομεακά τώρα, θέλουμε να κάνουμε κάτι για όλους. Εμείς όμως είναι απλό το μήνυμά μας Ο τρόπος όμως με τον οποίο λειτουργούν οι συμφωνίες για τις αεροπορικές υπηρεσίες είναι μοναδικός, δεν υπάρχει θέση αναδίπλωσης και γι' αυτό ελπίζω ότι καθώς μιλάτε με τους ομολόγους σας τα κράτη-μέλη σας μπορείτε να ενισχύσετε αυτή, το νόημα, αυτή την έννοια ότι πρέπει να εστιάσουμε στα αυτοκίνητα, στη φαρμακοβιομηχανία και αλλού, αλλά ότι οι αερομεταφορές έχουν διαφορετική φύση και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρόπ. 25 χρόνια εσωτερική αγορά είναι μια μοναδική ιστορία επιτυχίας για την αεροπλοεία. Θέλουμε να παραμείνει έτσι. Η Lufthansa στη Γερμανία ως ιδιωτική εταιρεία αγωνίζεται υπέρ των ανοιχτών αγορών κατά του προστατευτισμού και είμαστε στο πλευρό σας. Αν παραμείνει το Brexit θέλουμε να έχουμε μια συμπροματική ρύθμιση για τους ανοιχτούς ουρανούς και για εκείνους που συμμετέχουν στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να ισχύουν όλοι οι νόμοι που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να υπάρχει κοινωνία δύο κατηγοριών ή δύο ταχυτήτων. Έτσι μπορούμε να βρούμε γρήγορα μια καλή λύση. Δεν είμαι τελείως απεσιόδοξος. Μετά από μεγάλες διαπραγματεύσεις θα έχουμε μια ε, μεταβατική, μια επόμενη συμφωνία διάδοχη και μπορεί να αλλάξουν νόμοι και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει θαυμάσια ευκαιρία να παραμείνει. Είπαμε, για μια ελπίδα ζούμε. Και όπως είπε και ο κύριος Φαντεκάμπα ότι το Brexit είναι αδύνατο, μπορεί να καταλάβαμε σήμερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανατραπεί. Γιατί είπαμε, για μια ελπίδα ζούμε και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ο κύριος Πάστλαϊτνε. Ευχαριστώ πολύ σίγουρα το θέμα αυτό του Brexit είναι πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Εμείς λέμε να το δείτε με τρόπο ρεαλιστικό και τότε θα καταλάβετε ότι θα επηρεάσει τον τουρισμό και ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη των 27 με αρνητικό τρόπο αν δεν υπάρξει καμία συμφωνία, μια κακή συμφωνία για την αεροπορία. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Το σημερινό συμπέρασμα είναι ότι δεν επιτρέπεται να κλείσουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση. Το Κοινοβούλιο έπαιξε το ρόλο του, έδωσε βήμα ε, στους ενδιαφερόμενους, έγινε συζήτηση. Εγώ τι κρατάω. Αν έπρεπε να ψηφίσουν ε, όλοι οι παρόντες, όλοι θα ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακούσαμε τα θετικά της Ευρώπης, τα ερευνητικά προγράμματα, τον ενιαίο ουρανό, τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, το ρόλο του οργανισμού ΕΑΣΑ. Αυτά καθημερινά τα λέμε εμείς και θα πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το ευρωπαϊκό μοντέλο που βοήθησε για τη διαδρασιμότητα. Παρακαλώ ένα θερμό χειροκρότημα για όλο το πάνελ που τήρησαν οι ομιλητές τους χρόνους και μας ε, κοινοποίησαν τις θέσεις τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.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 Mes chers collègues, nous continuons. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τη συνεδρίασή μας, παρακαλώ. Si vous voulez discuter... Εάν θέλετε να συζητήσετε, σας παρακαλώ να συζητήσετε εκτός εθούσης. Έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε στην Επιτροπή μας τον κύριο Χέραλτ Withers κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής θα μάθουμε τα αποτελέσματα για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΜΗΕ, CEF δηλαδή στα αγγλικά, που υπήρξε αυτός ο τρίτος κύκλος ε, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, τρίτος κύκλος. Είχαμε ένα πολιετές πρόγραμμα και ένα ετήσιο πρόγραμμα. Στόχος είναι να καταργηθούν οι συμφορήσεις, αν θέλετε, τα, τα σημεία όπου υπάρχει τέλμα και να ενισχυθεί η σιδηροδρομική διαλειτουργικότητα, να βελτιωθεί το σχέδιο των μεταφορών το διασυνοριακό, Δεύτερος στόχος να εγγυηθούμε τα συστήματα μεταφορών τα οποία θα είναι αηφόρα, βιώσιμο, αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου για να προετοιμαστούμε για τις μεταφορικές ροές του μέλλοντος που προσδοκούμε να έχουμε και να βελτιώσουμε την ε, ένταξη, την ενοποίηση, τη διαλειτουργικότητα, την πολυτροπικότητα των ε, διαφόρων μορφών μεταφοράς, να επιτρέψουμε τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, του ανθρακικού αποτυπώματος και να έχουμε βελτίωση στις μεταφορές. Θα ήθελα να μάθω τα αποτελέσματα ε, και σας δίνω το λόγο κύριε Ρούτερς, Χαραλτ Ρούτερς. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είστε εδώ στο βήμα δίπλα μας, κοντά μας θα δείτε έναν άνθρωπο που δουλεύει πολύ σκληρά, που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για την Επιτροπή μας. Κάθε φορά που του ζητάμε κάτι είναι αμέσως ε, διαθέσιμος και με την καλύτερη δυνατή διάθεση. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που ε, είπατε όλα αυτά τα καλά λόγια για μένα. Είναι πραγματικά τιμή που εμφανίζομαι ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σας για να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα αυτής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντας. Θα σας ε, μιλήσω στα αγγλικά. Κυρίες και κύριοι, είχαμε τις προσκλήσεις του 2016 CEF και θέλω να αναφερθώ και ε, στις δηλώσεις της Επιτρόπου όπου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ε, είχαμε υπερβολική εκδήλωση ενδιαφέροντος, πάρα πολλοί απαντώντες, έχει ήδη αναφερθεί το χρονοδιάγραμμα. Εγώ θα σας, δώσω κάποια σύντομα αποτελέσματα εν συντομία. Έγινε συζήτηση σήμερα το πρωί και με την Εστονή Υπουργό και με την Αρμόδια Επίτροπο, οπότε τα ξέρετε τα περισσότερα δόθηκε έμφαση στο εργαλείο Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη αλλά και στην ψηφιακή αγορά, στην ψηφιακή εποχή. Να τονίσω ότι είναι τρίτος κύκλος, τρίτη επιλογή. Έχουμε επενδύσεις 2,7 δις και ολοκληρώνεται ένας κύκλος τριών προσκλήσεων εκδήλωση ενδιαφέροντος το 14, 15 και 16. Ήταν μια δέσμευση που είχαμε υιοθετήσει με τις χώρες της Βαλτικής κυρίως με τις χώρες που εντάσσονται στο Ταμείο Συνοχής ε, γιατί είχαν εξαντλήσει τους δικούς τους χρηματοδοτικούς φακέλους. Κάποια βασικά μηνύματα σε δύο διαφάνειες πριν προχωρήσω σε λεπτομέρειες. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση, 3,8 φορές συνολικά καλύφθηκε ε, με προσφορές και 6,5 φορές ε, καλύφθηκε ε, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το φάκελο συνοχής. Ουσιαστικά μιλούμε για 11,3 δι του φακέλου για τη συνοχή και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Πρέπει να σημειωθεί από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ. Κανεί δεν το περίμενε αυτή η μεταφορά των 11,3 δις από το φάκελο της συνοχής να πάει στο εργαλείο Connecting Europe συνδέοντας την Ευρώπη και να είναι τόσο επιτυχημένη και να επιτρέπει να απορρόφησε 11,3 δις μέσα σε τρία χρόνια. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλω να πάρετε. Και Βλέπετε στην τελευταία παράγραφο ότι αυτό σημαίνει ότι μοιραζόμαστε τα χρήματα, δηλαδή όλοι αξιοποιούν πλήρως τους φακέλους τους, αλλά έχουν ήδη μπει και στη φάση της εφαρμογής της υλοποίησης 640 εκατομμύρια ε, ήρθαν πίσω για επανέγχυση αν θέλετε ε, re-injection. Να σας δώσω ένα παράδειγμα με, τις, ε, με τους διαγωνισμούς το 14-15 και στις αρχές του 16 οι συμμετέχοντες ήταν ήδη ικανοί να εξοικονομήσουν 500 εκατομμύρια και τα οποία ξαναμπήκαν στο, στο διαγωνισμό και μπορούσαν να επιλεγούν και άλλα δύο έργα. Ένας πολύ επιτυχημένος τρόπος δηλαδή να εφαρμόζουμε, να υλοποιούμε τα έργα που από κοινού επιλέγουμε. Ένα άλλο βασικό μήνυμα που θέλω να στείλω με αυτή μου την παρέμβαση εδώ στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αυτό που έχει να κάνει με το αίτημά σας, κυρία Πρόεδρε. Χρήματα να μην πάνε μόνο στα μεγάλα έργα, αλλά και στα μικρότερα διασυνοριακά για να καλυφθούν οι αδύναμοι κρίκοι. Είχαμε συμφωνήσει ότι 140 εκατομμύρια θα τεθούν κατά μέρο για μικρού μεγέθους διασυνοριακά έργα. Και εδώ είχαμε υπερπλήρωση και υπερκάλυψη ε, στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έχουμε υπερβολική ευελιξία, 20% ε, παραπάνω ε, υπέβαλαν προτάσεις. Επιλέξαμε 13 έργα που έχουν περάσει με επιτυχία το στάδιο της ε, εξωτερικής αξιολόγησης και το ύψος του προϋπολογισμού είναι 140 εκατομμύρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Άρα για τα έτη 14, 15 και 16 έχουμε 604 έργα που επιλέξαμε, 2.000 θα είναι περίπου και όχι, Έχουμε συγχρηματοδότηση 21,4 δις ευρώ για το Connecting Europe Facility, πάνω από το 90% του συνολικού προϋπολογισμού των ενισχύσεων και συνολική επένδυση 41,6 δις ευρώ. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τους στόχους. Δεν θα μακρηγορήσω στόχος λοιπόν ήταν τριπλός το 2016. Πρώτον, να γεφυρώσουμε ε, τα χάσματα, να καλύψουμε, να ενισχύσουμε τους αδύναμους κρίκους, να αφαιρέσουμε τα σημεία στο οποίο υπάρχει τέλμα, να ενισχύσουμε την αηφορία, την αποτελεσματική μεταφορά σε βάθος χρόνου, να βελτιώσουμε την διασύνδεση, την συνδεσιμότητα, την διαλειτουργικότητα, και ο προϋπολογισμός μοιράζεται ε, σε αυτούς τους τρεις στόχους, για να επιτευχθούν και οι τρεις αναλόγως. Εδώ βλέπετε τα αιτήματα χρηματοδότησης ύψους 7,5 δις ευρώ σε 332 έργα. Οι εξωτερικοί αξιολογητές μείωσαν αυτά τα αιτήματα σε 5,5 δις ευρώ και σε 208 έργα και πρέπει αυτά να συγκριθούν με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό που είναι σε μπορδό και κόκκινο 2,5 ε, δις ευρώ και 639 έργα και βελτιώσαμε τις δυνατότητες με ευελιξία 20% και τελικά έχουμε προϋπολογισμό 2,659 δις ευρώ και 152 έργα. Χρειάστηκε λοιπόν να μειώσουμε σημαντικά από το πορτοκαλί στο πράσινο. Περικόψαμε πολλά έργα τα οποία εγκρίνουμε αλλά για τα οποία δεν έχουμε χρήματα. Δυστυχώς. Εδώ βλέπετε την κατανομή των χρημάτων αναφάκελο, αναστόχο. Για παράδειγμα, έχουμε υπερβολική εκδήλωση ενδιαφέροντος για το στόχο της συνοχής και είναι τεράστιο η προσπάθεια συγχρηματοδότησης ύψους 1,7 δις ευρώ. Πολύ λίγα χρήματα από τις χώρες συνοχής πηγαίνουν στο ετήσιο πρόγραμμα, ενώ για το πολιετές πρόγραμμα καταβάλουμε προσπάθειες να είναι περισσότερα τα διαθέσιμα χρήματα, γενικότερα για το ETMS, για την καινοτομία και το καθεξής και το ετήσιο προ... πρόγραμμα βλέπετε και τα μικρά έργα αλλά χαρακτήρα. Με περισσότερες λεπτομέρειες θα δούμε πού πάνε τα, τα χρήματα σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια τώρα, την επόμενη διαφάνεια. Σας βοηθώ γιατί είναι πολύ μικρά τα γράμματα στην οθόνη. Η αριστερή στήλη πιο μεγάλη είναι για τους βασικούς διαδρόμους του δικτύου. 1,265 ε, δις και 297 εκατομμύρια για το ERTMS. Και ε, το δεύτερο από αριστερά είναι άλλα τμήματα του βασικού διαδρόμου, το τρίτο από αριστερά η σιδηροδρομική διαλειτουργικότητα, το πέμπτο από αριστερά η καινοτομία και το καθεξής. Εδώ βλέπουμε με κόκκινες στήλες το γενικότερο φάκελο σε εκατομμύρια ευρώ. Μεγαλύτερος φάκελος είναι το ΣΕΣΑΡ, ΣΕΖΑΡ, μετά, ε, τρίτο από αριστερά, πρώτος από αριστερά ERTMS, δεύτερο από αριστερά καινοτομία, τέταρτο από αριστερά ITS και έχουμε τέταρτο από δεξιά έργα για το βασικό δίκτυο και τα συνολικά δίκτυα, Core και Comprehensive Networks. Ως προς τις προτεραιότητες, το γενικότερο μήνυμα είναι ότι ε, έχει υπερκαλυφθεί αυτή η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο. Έχουμε βελτιώσει τον προπολογισμό όσο περισσότερο μπορούμε. Οι πόροι του Ταμείου Συνοχή έχουν αξιοποιηθεί μέχρι το τελευταία δεκάρα και θα έχουμε πρόσθετο προπολογισμό για τα μικρά διασυνοριακά έργα. Αυτό είναι σημαντικό. Είδατε αυτό το τεύχο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλου εσά. Είναι η τρίτη λευκή βίβλος τούβλο που έχει δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια. Μετά από αυτό θα μείνει κάτι λιγότερο από ένα δις για τα χρόνια 18, 19 και 20. Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε, θα συνεργαστούμε με τα μέλη της Κοινοβουλευτική Επιτροπής σας για την πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων. Πάντοτε κανείς πρέπει να το χρησιμοποιεί, αλλιώς θα το χάσει. Είναι γνωστός ο κανόνας και θέλουμε αυτά να συνεχιστούν το 18, το 19, το 20 και θα επανέλθουμε στην Επιτροπή σας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τελευταία άσκηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσφορών και το καθεξής. Σας ευχαριστώ θερμά. Ε, κυρία Πρόεδρε, για τα αποτελέσματα, για τη δουλειά σας. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με τη συνεργασία που έχουμε με εσάς, με τα λοιπά μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με τα κράτη-μέλη, ειδικότερα για το εργαλείο για τη διασύνδεση στην Ευρώπη. Δείχνουμε, δείχνουν όλοι ότι είναι ικανοί να, να, να απορροφήσουν τον υφιστάμενο προϋπολογισμό, να δώσουν προτεραιότητα ε, στα εναλλακτικά καύσιμα, σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, στην καινοτομία, στα διασυνοριακά έργα τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία ε, για τα συνολικά δίκτυα μεταφορών. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως για την ύπαρξη αυτής της συνεργασίας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια ε, στις εργασίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρέτερς για τη σαφήνεια αυτή και το δυναμισμό σας. Ε, σας διακρίνει γιατί σας βλέπουμε συχνά εδώ και το ξέρω. Ο Βιμ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεταδοτικός ο ενθουσιασμός του κυρίου Ρόιτερς μετά από αυτό το δύσκολο απόγευμα που είχαμε για το Brexit, καλό είναι να ακούμε και κανένα θετικό. Να έχουμε μια ένεση θετική, ε, στο και αν είναι δισεκατομμύρια ευρώ αυτά. Αλλά έχω μπερδευτεί με τα νούμερα και έχω και κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, θα πάρω αυτή τη βίβλο στις διακοπές μου, αυτό το τούβλο να το μελετήσω στις διακοπές και να το συγκρίνω και με άλλες βίβλους, μήπως έχουμε τίποτα λάθη και τίποτα επικαλύψεις ως προς τα νούμερα. Όχι, δύο ερωτήσεις έχω όμως. Πρώτον, ο ρυθμός των εκταμιεύσεων, των πληρωμών, τι λέει ο κύριος Ράιτερς, ότι είμαστε στο παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο λύγει 31 Δεκάτου του 2020. Είναι εξασφαλισμένες οι εκροές. Μην έρθουμε ένα χρόνο αργότερα. Δύο ερωτήσεις έχω λοιπόν πώς έχει ο ρυθμός των εκταμιεύσεων, γιατί μπορεί να χρειαστεί άλλος ένας χρόνος για να αποφασίσουμε το νέο PDP. Γιατί θα έχουμε τις ευρωεκλογέ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Χωρίς να θέλω εγώ να προκαλέσω κανένα πρόβλημα. Δεύτερη ερώτηση. Η Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειακής Πολιτικής τι μαθαίνει από την επιτυχία αυτή. Έχουμε τα χρήματα από την συνοχή και τα αξιοποιούμε. Συνεργάζεστε τώρα καλύτερα με τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο. Σας φθονούν, σας ζηλεύουν, σας ε, βάζουν τρικλοποδιές. Και τι λένε για τα κονδύλια. Α, τα παίρνουμε από την ε, συνοχή, δεν το ήξερα. Ε, και τελευταία ερώτηση. Η θέση της Γενικής Διεύθυνσης MOVE είναι ενισχυμένη απέναντι στον Ότιγκερ. Και σας έχουμε καλή επιτυχία κύριε Reuters. Αλλά να το αξιοποιήσει η κυρία Μπούλς για να είναι εγγυημένο το συνδέοντα στην Ευρώπη, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το blending, ο συνδυασμό χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Κύριε Γιάννα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου ε, τον κύριο Ρετές για την εργασία του που μπόρεσε να φτάσει από, να, να απαντήσει σε όλα αυτά τα αιτήματα που προέρχονται από κάθε γωνία και από την κάθε μας περιφέρεια. Εγώ είμαι λοιπόν πολύ ευχαριστημένη και ήθελα να διαβιβάσω τη χαρά μου και τη συγκίνησή μου γιατί βρήκαμε το κρίκο που έλειπε από την αλυσίδα γιατί έτσι έχουμε αυτές τις μελέτες, έχουμε την οριστική μελέτη και βεβαίως εφόσον πρόκειται για μια κοινή εργασία με τις δυο περιφέρειες, έτσι το είδαμε και ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά αυτό που θα ήθελα επίσης είναι, όπως είπε και ο κύριος Βαντρικάμπ και το τόνισε, Αρχίζουμε να κάνουμε πετάλι, να προσπαθούμε για να μπορέσουμε να καταφέρουμε επόμενος προπολογισμό για τις υποδομές μας να σταθεί στο ύψος των φιλοδοξιών που εμείς ήδη έχουμε υποβάλει. Έχουμε υποβάλει όχι μόνο το αίτημα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή οι υπηρεσίες σας να αρχίσουν να υπολογίζουν πόσα χρειάζονται ώστε να ολοκληρωθούν οι δεσμεύσεις που μας παρουσιάσατε το 2014, 2015 και 2016 και τα όσα έπονται. Να έχουμε δηλαδή ένα τρόπο να υπολογίσουμε, να έχουμε ένα πρώτο νούμερο. Τι χρειάζεται σε σχέση με τις δεσμεύσεις που, και τις υποχρεώσεις που ήδη έχουμε. Το δεύτερο το είπατε και εσείς ο ίδιος, τα αιτήματα όσα μας ζήτησαν και πόσα δεν μπορέσαμε να δώσουμε. Ένα μεγάλο αριθμό που ήδη φαίνεται και να δούμε ποιο είναι το ρεαλιστικό κομμάτι πάνω στο οποίο δουλεύουν οι υπηρεσίες σας. Έπειτα έχουμε και το θέμα της μεθοδολογίας. Πιστεύω πως αυτή η στάση, η μεθοδολογία ΣΕΦ, θα πρέπει να την παρουσιάσουμε όχι τόσο για να την ε, υποβάλουμε και στην ε, Ρέτζη, αλλά και γιατί εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να τονίσουμε τις επιτυχίες, να δούμε δηλαδή και να συνομιλήσουμε με όλους μας τους συνομιλητές αυτής της γραμμής, να τους πούμε ότι γιατί έτσι μπορέσαμε και πρέπει να τις επιβάλλουμε και στην, στην ε, ΕΤΕΠ ώστε να ε, δούνε ακριβώς πώς έχει λειτουργήσει αυτή η, ε, η μεθοδολογία. Και όχι μόνο βοηθάει, όπως εσείς ο ίδιος το είπατε, στις χώρες της συνοχής, ώστε να επενδύσουν καλύτερα και να βελτιώσουν και την ποιότητα των επενδύσεών τους, με τρόπο μάλιστα πολύ πιο απαιτητικό και ποιοτικό, αλλά βοηθάει και γιατί δίνει τρόπους στα δεξιά και στην αριστερά, δηλαδή το κομμάτι Rage Ε, και εκείνους τους πιο καινοτόμους εντός εισαγωγικών που είναι το ΕΦΣΙ, το η ΕΤΕΠ e και τα λοιπά, ώστε να μπορέσουν όλα αυτά να μπουν, να δρομολογηθούν, να αρχίσουν να κινούνται, όπως είπατε, με τον εκτελεστικό οργανισμό που πλέον έχουμε πολλή δουλειά λοιπόν και σας στηρίζουμε και θα σας στηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σέντερ και ο κύριος Κράμερ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ κόπος από πίσω, δεν το διάβασα ακόμα ολόκληρο. Μερικές προφορίες τις κοίτασα. Γιατί μου είπε ο Βιμ Βαντεγκάμπ, πρέπει να αναφέρω τους κρίκους που λείπουν, έχουν γίνει πολλά, 110 εκατομμύρια έχουμε και υπερπροσφορά. Είναι καλό γιατί συνεργαστήκαμε και με την Επιτροπή των Περιφερειών. Και είναι σημαντικό το θέμα και αυτό ε, συνενώνει την Ευρώπη. Απλώ θα επιθυμούσα να είχαν γίνει αυτά πριν από 30 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα, κάλιο αργά παρά ποτέ. Έχω δύο ερωτήσεις. 40%, 40 εκατομμύρια πηγαίνουν μέχρι τα σύνορα στην Ανατολική Γερμανία και την Πολωνία προς το Βρότσλαβ και κλείνει το μικρόφωνο. Έχετε διαπραγματευτεί με την Ομοσπονδική Κυβέρνηση Γερμανίας να το κάνω αυτό την άλλη φορά που λείπει, γιατί ακούω ότι το κρατήδιο του Βραδεμβούργου ήθελε να κάνει το σχεδιασμό για αυτή τη διαδρομή να το προχρηματοδοτήσει και το απαγόρευσε ο Υπουργό Μεταφορών της Γερμανίας γιατί προέχει το Ομοσπονδιακό Σχέδιο. Εδώ έχουμε ένα ευρωπαϊκό έργο πολύ σημαντικό δεν θέλει καμία σχέση να έχει η γερμανική την κυβέρνηση, κοιτάει μόνο το εθνικό της πλάνο. Ε, πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση για να το καταλάβει η γερμανική κυβέρνηση και την άλλη φορά να χρηματοδοτήσει τη διαδρομή, ε, τη χαραξη κότπου Κότπους-Χόρκα. Για τον αυτοκινητόδρομο υπάρχουν τώρα κάποιες χώρες που δεν έχουν καθόλου διόδια. 100% έχουν, με βάλει διόδια στο σιδηρόδρομο και 1% στους αυτοκινητοδρόμους. Πώς γίνεται εκεί η χρηματοδότηση, υπάρχουν κάποια κριτήρια, σε ποιο ύψος χρηματοδοτούνται. Αυτοκινητόδρομοι με ή χωρίς διόδια. Σε κάθε σιδηρόδρομο και σε κάθε έργο βάζουμε τέλη. Στην Τσεχία είχαμε προβλήματα στους αυτοκινητοδρόμους, έτσι έμαθα. Άκουσα να λέει, είπε λέει ο κύριος Γιούνκερ ότι θα το εγκρίνει. Ε, χωρίς να ληφθούν υπόψη όλες οι ρυθμίσεις ή να τηρούνται. Θα υπάρξει ε, ε, συγχρηματοδότηση ε, ακόμα και όταν δεν κάνουμε μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου στην Τσεχία, γιατί κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Ευχαριστώ, κύριος Μάρκος Πίπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση. Το υπενήχθη ο κύριος Βαντενκάμπ. Οι χώρες της συνοχής δήλωσαν ότι έχουν προβλήματα για το ΣΕΦ, ε, το Connecting Europe Facility. Δεν ήταν πολύ εύκολο να γίνει διαπραγμάτευση. Πώς γίνεται τώρα η κατανομή των πόρων. Υπάρχουν κάποιοι φάκελοι, εθνικά κονδύλια, ε, κάποια κράτη ε, προτιμούνται, κάποιοι δεν συμμετέχουν. Υπάρχει κανένας χαμένος, υπάρχει καμιά χώρα που να μην έχει καθόλου έργα. Και εδώ συνδέεται με το προηγούμενο το ερώτημά μου. Τελικά πώς βλέπετε το μέλλον του Connecting Europe. Θα υπάρξουν κάποια χρήματα που δεν θα απορροφηθούν, γιατί στο παρελθόν το είχαμε δει σε περίπτωση που δεν είχαν απορροφηθεί όλα τα κονδύλια. Ε, μπορούσαν όλες οι περιφέρειες να υποβάλουν υποψηφιότητα για να τα ανακτήσουν σε περίπτωση μη εξάντλησης των πόρων. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πίπερ. Ο κύριος Κούν τελευταίος. Merci, Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για το αποτέλεσμα που μας παρουσιάσατε κύριε Ρόιτερ. Γιατί ο συνδυασμός Connecting Europe Facility και κονδύλια από τα περιφερειακά και τη συνοχή, κατά την άποψή μου είναι απολύτως και τρομερά σημαντικός για να έχουμε η ανάπτυξη της οικονομίας και βελτίωση της κατάστασης, ιδιαίτερα στην ανεργία των νέων. Ακριβώς στις χώρες αυτές, όπου έχουμε μεγάλες ανησυχίες. Είναι χώρες που έχουν αδυναμίες ε, στις υποδομές τους και στις διορθωτικά ταμεία. Στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία βλέπω με χαρά και στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία και στην Πορτογαλία και στην Ιταλία, Νότια Ιταλία. Σημαντικά τμήματα των διευρωπαϊκών αξώνων και δικτύων. Αυτό έχουν και υψηλή προστιθέμενη αξία για την κυκλοφορία και βελτιώνουν τους άξονες. Αυτές είναι υποδομές κοντά στην οικονομία και μόνο έτσι θα δώσουμε μια πρώτη όθηση σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να ε, μπαίνουν και οι δημόσιες προμήθειες εκεί που είναι το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της οικονομίας. Το δεύτερο είναι να πάνε να εγκατασταθούν επιχειρήσεις σε αυτές τις περιφέρειες. Έχουμε κάνει πολλή συζήτηση, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και κανένας δεν ήθελε ένα blending ή μείγμα από το δικό του ταμείο. Όλοι ήθελαν να τα κρατήσουν στο δικό τους έλεγχο το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το, ήθελα να το κρατήσουν οπωσδήποτε ε, ε, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών. Εμείς θέλαμε το ΣΕΦ και μην το ακουμπήσει κανένας. Τώρα βλέπουμε ότι πήραμε τη σωστή απόφαση. Και σε αυτό το δρόμο θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Και διάβεσα στη Γερμανία, στη Wirtschaftswoche, ένα ωραίο άρθρο, η Ευρώπη ανακάμπτει, ανακάμπτει οικονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. 3,5% φέτος και του χρόνου θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Και ακριβώς στις χώρες που το χρειάζονται περισσότερα και συμμετέχουν και αποφελούνται, ε, είναι η σωστή φιλοσοφία. ερωτήσει δεν έχω. Πού να έχω. Ε, ευχαριστώ κύριε Κούν. Εγώ είχα δύο μικρές ερωτήσεις. Η πρώτη αναφέρεται στην ακρόαση ότι με το Brexit τι θα γίνει για τα project που έχουν χρηματοδοτηθεί και θα βγουν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα συνεχιστούν. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερο που θέλω να ξέρω είναι αν μια χώρα που έχει βάλει project στο μηχανισμό διασύνδεσης και λόγω αλλαγής κυβέρνησης μετά από εκλογέ, χωρί να οικογένειε ονόματα δεν λέμε, οικογένειε δεν φύγουμε μπορεί να επανέλθει. Ποια είναι η διαδικασία το κράτος πρέπει να αποζημιώσει τα χρήματα που έχει καταβάλει ήδη η Ευρώπη. Τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση. Ευχαριστώ κύριε Ρόιτρες. Εκ των προτέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ συνάδελφοι για τις ερωτήσεις. Πολλές από τις ερωτήσεις αφορούσαν χώρες συνοχής και τον προπολογισμό της συνοχής βέβαια. Αυτός ο προπολογισμό της συνοχής που μπήκε στο ε, ε, διευκόλυνση για τη σύνδεση της Ευρώπης αφορά τις χώρες ε, συνοχής και η συμφωνία που προέκυψε από εδώ ήταν να χορηγηθούν στη διάρκεια τριών ετών σύμφωνα με τα εθνικά κονδύλια και είχαμε κάνει τρεις προκηρύξεις ε, για αυτές τις χώρες ώστε να καταναλώσουν τον εθνικό τους κονδύλιο. Ας πούμε από τα 11,3 δις, 4 δις για την Πολωνία και η Πολωνία είχε τρεις φορές τη δυνατότητα να μας υποβάλει ε, projects για να καταναλώσει αυτά τα χρήματα. Και η Πολωνία μπόρεσε, όπως και οι υπόλοιπε χώρες, συνεχίζουν να το κάνουν αυτό και να τα καταναλώσουν και να τα καταναλώσουν και τελείω τα κονδυλιά τους, γιατί είχαμε και παραπανήσια ε, project, 6-7 φορές παραπάνω κονδύλια. Η ανάλυση που κάνουμε είναι ότι αυτό οφείλεται στα στοιχεία στο στοιχείο του ανταγωνισμού, ότι πλέον μετά τα τρία χρόνια τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να πάνε μόνο για μία χώρα συγκεκριμένη, αλλά ότι μεταξύ τους οι χώρες θα πρέπει να ανταγωνιστούν. Υπήρξε μια χώρα, ας πούμε, θα δείτε στο τέσσερις χώρες που δεν κατανάλωσαν αρκετά τα χρήματα. τα χρήματα που δεν καταναλώθηκαν ήταν 17 εκατομμύρια. 70, συγγνώμη, 7, 0, 70 από τα 11,3 δις. Ελάχιστα δηλαδή, ήταν λιγότερο από 1%, ήταν 0,0 κάτι σε σχέση με όλο τον προπολογισμό. Τα χρήματα που δεν απορροφήθηκαν ήταν πολύ λίγα, δεν ήταν σχεδόν δυνατόν το δίκανη. Αν θέλει πρέπει πραγματικά να το ψάξει αυτό το φυλάδιο. Αυτά τα 70 λοιπόν εκατομμύρια πώ κατανεμήθηκαν. Τα κατανείμαμε με βάση τι αρχέ του ΣΕΒ, καταρχάς ευρωπαϊκά project, δηλαδή διασυνοριακά, με διασυνοριακή διάσταση, και εκεί δόθηκαν αυτά τα χρήματα, δηλαδή ε, η οδός Βαλτική και τα λοιπά, μια ένα δυσυνορικό project της πολωνο-τσεχικό και ένα Σλοβενικό. Αυτά. Και έτσι απορροφήθηκαν και αυτά τα 70 εκατομμυριάκια. Πολύ μικρό ποσό, και έτσι λοιπόν πολύ επιτυχώς εφαρμόστηκαν όλα αυτά και αν κάτι μας δάσκει αυτό, μας διδάσκει ότι τα χρήματα της συνοχής με λίγο συναγωνισμό, με λίγη άμυλα, ευγενή, μπορεί να μπορούν να απορροφηθούν όλα αυτά τα κονδύλια. Ήδη από την αρχή της περίοδου και με χαρά είδαμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα των χωρών της συνοχής και όπως είπε και ο κύριος Κούν είναι καλά για project τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας. Και αυτή είναι και η παραπληρωματικότητα που έχουμε στην DG Radio, γιατί βασικά κάνουμε διασυνοριακούς σιδηροδρόμους και μετά οι, συν, συνάδελφοι της συνοχής στη Radio κάνουν τα άλλα κομμάτια. Ας πούμε, εμείς κάνουμε σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ ε, Βαρσοβίας και Λιθουανίας και, και η Regio κάνει τα υπόλοιπα. Και επειδή έχουμε Ε, μπορούμε να δώσουμε πέντε φορές παραπάνω σε αυτούς για τα project που δεν έχουμε μπορέσει να χρηματοδοτήσουμε. Ο κύριος Κράμερε πολύ συγκεκριμένα ρώτησε Χόρκα ε, χρήματα έχουν δοθεί αλλά βεβαίως με τον διάλογο που έχουμε, το θετικό διάλογο που έχουμε, θα τονίσουμε, ξέρετε και εσείς ότι συζητάμε με την ε, Βερανδεβούργο και με άλλα κρατήδια, δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι, αλλά ολόκληρη η σύνδεση αυτή και σίγουρα μαζί με εσά και άλλους θα ε, δραστηριοποιηθούμε εκεί και Όσον αφορά τι οδικές μεταφορές, οι οδικές μεταφορές ήμασταν πολύ περιορισμένοι. Μιλάμε για ασφαλή ε, χώρους ε, στάθμευσης. Δεν κάνουμε εθνικά τμήματα. Οι χρήματα που πάνε στου δρόμου. είναι πολύ λίγα και αν υπάρχουν εθνικά project που πρέπει να, να, να, να γίνουν, το κάνουμε μέσω του ΕΦΣΥ. Και μετά έρχεται και το θέμα σας για τα διόδια. Ε, στα, στα ΕΦΣΙ χρειάζεται και συγχρηματοδότηση, ως εκ τούτου βάζουν και διόδια σε αυτούς τους δρόμους. Τώρα, για την αλλαγή, πιθανή αλλαγή κυβέρνησης. Για το Brexit, για την ώρα τα project με το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζονται, είναι υπό εκτέλεση, γιατί για την ώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν υπάρχει αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων. Οπότε τα project που έχουμε από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εύκολο να τα διαχειριστούμε, γιατί τα περισσότερα εξ αυτών θα ολοκληρωθούν το 2019, οπότε θα είναι σχετικά απλό. Αυτή είναι η κατάσταση. Βεβαίω θα υπάρξει μια λεπτομερή ανάλυση τη στιγμή που θα λάβουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορώ εκ των προτέρων εγώ να πάρω θέση. Τώρα, για την ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνηση, βεβαίω υπάρχουν αλλαγέ κυβέρνηση παντού και όλη την ώρα. Αυτό δεν αλλάζει απαραίτητο στι δεσμεύσει τι δικέ μα με την εκάστοτε κυβέρνηση μέσω της σύναψης συμφωνιών χρηματοδότησης που έχουμε. Εάν μια συμφωνία χρηματοδότησης δεν γίνεται σεβαστή γιατί το κράτο μέλο δεν σέβεται το δικό του κομμάτι τη συμφωνία, τότε δεν απορροφάται ο προπολογισμό και επανέρχεται σε εμά. Γιατί υπάρχει ο μηχανισμός use it or lose it. Ή θα το χρησιμοποίησει ή θα το χάσει. και τότε τα χρήματα αυτά ξαναμπαίνουν στον ανταγωνισμό μέσω στον συναγωνισμό μέσω τη προκήρυξη υποβολή προσφορών. Υπήρχε και η ερώτηση του κ. Βαντρικάμπα για το ρυθμό των πληρωμών και τον ένα, 1 ίσιν δύο. Ίσως ο Ανδρέας Μπός που είναι επικεφαλής του τμήματος ε, να μπορέσει να απαντήσει. Πρόεδρε, μάλιστα. Ξεχάσετε και τη δική μου ερώτηση για την Τσεχία και τον αυτοκινητόδρομο. Με την άδειά σας θα προσπαθήσω να απαντήσω και στι δύο ερωτήσεις του κυρίου, και του κυρίου Βανταγκράπ και του κυρίου ε, Κράμερ. Είμαι επικεφάλη τμήματάρχη ε, για αυτό το θέμα, για τι μεταφορές ενέργειας και τεχνολογίες τη ε, Προσπαθούμε να έχουμε ε, κοινή ε, διαχείριση. Για τον κύκλο των πληρωμών, χωρίς να μπω σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, θέλω να σας ε, βεβαιώσω ότι είναι σφιχτός ο διαχειρισμός. Έχουμε δόσεις πολυετής από την ανάληψη υποχρεώσεων. Έχουμε ανάληψη υποχρεώσεων για συγκεκριμένο έτος βάσει των αναγκών ε, του έργου και για τις πληρωμές έχουμε μια πρώτη προκαταβολή, μια ενδιάμεση προκαταβολή πάντα βάσει των αναγκών του έργου, τι πραγματικά χρειάζεται και μετά κάνουμε την εξόφληση ε, με βάση το κόστος έτσι ώστε να έχουμε μια κανονική ροή πληρωμών, μια κανονική εκταμίευση και να υπάρχει αρκετή ρευστότητα ανα πάσα στιγμή για να συνεχίσετε το έργο. Απ' την άλλη μεριά δεν θέλουμε κάπου να παραμένουν τα χρήματα και να αποτελματώνονται, γι' αυτό δεν δίνουμε πάρα πολλά σε κάθε δόση. Προσπαθούμε και σε στενή συνεργασία με τους δικαιούχους να τα καλύπτουμε αυτά. Απαντώ στον κύριο Κράμαρα, μου επιτρέπετε, για τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, γενικότερα ε, ίσως στην επιλογή και την αξιολόγηση. Οι συνάδελφοι της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος συμμετέχουν πλήρως και τσεκάρουν αν ε, ε, προσαρμόζεται και συμμορφούνται πλήρως στο έργο με την περιβαλλοντική ε, νομοθεσία υπάρχουν αιρεσιμότητες, όροι και συνθήκες και στη Συμφωνία για την Εκταμείευση και πάντα το βλέπουμε αυτό σε συνεργασία με τους συναδέλφους Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και φροντίζουμε πάντα να συμμορφώνονται και διασταυρώνουμε με τους συναδέλφους αυτούς ε, τα ορόσημα και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ε, δρακόντια ελέγχει αυτά τα θέματα ε, συμβατότητας, πώς, θα λένε αυτά τα, διαδικαστικά ε, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αντικτύπου κτλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε πολύ τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών μου ε, που βρίσκει το χρόνο και έρχεται να μα εξηγεί όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Αξίζεται ένα χειροκρότημα. Tandis euh, ε, τώρα τελειώσαμε για σήμερα τις εργασίες μας. Όσους δεν σας ξαναδώ, ραντεβού 31 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί όμως. Για τους υπολείπους, θα σας δω την άλλη εβδομάδα στη Σουηδία που έχουμε αποστολή, διότι ε, οι εργασίες μας συνεχίζονται ακόμα και στις αντιπροσωπείες. Καλές διακοπές, καλή σας ξεκούραση, ευχαριστούμε κύριοι, κύριες διερμηνείς που μας θυμάται με την παρουσία σας, τον επαγγελματισμό σας, καλές διακοπές, καλές διακοπές, ξεκουραστείτε όλοι και δυναμικά να επανέλθετε γιατί μας περιμένει πολλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την